So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε αν θέλετε. με το απογευματινό μας πρόγραμμα και το 25 το σχέδιο εκθέσεως για τη μη συνέχιση των, ε, της αλλαγής ώρας της εποχιακής αλλαγής ώρας. Δεν πρόκειται για νέο φάκελο στη Γιούρη. Είχαμε δημόσια διαβούλευση το 2015. Η πρακτική της αλλαγής της ώρας ενεγράφει στην ενωσιακή νομοθεσία για δεκαετίες αλλά ανέκυψαν αντιδράσεις και διαφωνίες ενώσεων πολιτών, οι οποίες εκφράστηκαν όχι μόνο στη δημόσια διαβούλευση, αλλά και μέσω διαφόρων πρωτοβουλειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο οδήγησε σε ερωτήματα προς την Επιτροπή επ' αυτού, εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν πέρσι το Φεβρουάριο σε ψήφισμα του Κοινοβουλίου στο οποίο ζητούμε από την Κομισιόν να προχωρήσει σε πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου και αν κριθεί απαραίτητο πρόταση αναθεώρησης. Δημοσίευσε το καλοκαίρι η Κομισιόν τα πορίσματα μιας διαβούλευσης με 40 1,6 εκατομμύρια απαντήσεων που ήταν το μεγαλύτερο μέγεθος που είχαμε λάβει σε οποιαδήποτε δημόσια δεμούλευση της Κομισιόν. Έσπασε το ρεκόρ κατά 9 φορές το προηγούμενο ρεκόρ. ζητώντας να καταργηθούν οι εποχιακές αλλαγές της ώρας Αποτέλεσμα τούτου ήταν ότι ο πρόεδρος Κομισιόν Juncker στο State of the Union πέρυσι ενημέρωσε ότι η Κομισιόν επεξεργαζόταν οδηγία η οποία θα τερμάτιζε τις εποχιακές αλλαγές της ώρας με βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα το ενισχύ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση από τα κράτη-μέλη τα οποία από εκεί πέρα θα ήταν ελεύθερα να επιλέξουν την ώρα που θα ίσχυε στο, στην επικράτειά τους. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών από την εισηγήτρια κυρία Ούλσκοκ δίνουν περισσότερο χρόνο προσαρμογή στα κράτη-μέλη. Η οδηγία είναι να τεθεί ενισχύ από τον Απρίλιο φέτος με τελευταία αλλαγή ώρας τον Οκτώβριο όπως θα πρότεινε η Κομισιόν και δύο έτη προθεσμία με την γραφή για τα κράτη-μέλη διανεμήθηκε και το σχέδιο γνωμοδότησης την περισμένη εβδομάδα επί του θέματος αυτού με συνθήκες και προϋποθέσεις σε διάφορες περιφέρειες και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία θα πρέπει πάντως με συντονισμένο τρόπο να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί, αλλά θα ήθελα να κάνω μία-δύο ακόμα διευκρινήσεις επί του φακελού αυτού. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι οι εποχιακές αλλαγές της ώρας δεν επηρεάζουν μόνο την λειτουργία της ιστορικής αγοράς, αλλά έχουν διαστάσεις προστασίας δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα ως προς μειοψηφούσες ομάδες του πληθυσμού, επί των οποίων υπάρχει δυσανάλογος αντίκτυπος από τον κύκλο αλλαγής της ώρας. Ο, άθρο, αριθμός των ατυχημάτων και καρδιακών επεισοδίων φαίνεται ότι έχει αυξηθεί σε σχέση με την αλλαγή αυτή και προτείνω να συμπεριληφθεί παραπομπή στις μελέτες αυτές. Επίσης, τα θεσμικά όργανα στην Διαθεσιμική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία έχουν δεσμευτεί ως προς το ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου είναι ουσιαστικά εργαλεία για την βελτίωση της ενωσιακής νομοθεσίας και επομένως είναι ατυχές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε σχετική αξιολόγηση αντικτύπου ούτε σε διαβούλευση 12 εβδομάδων όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Ιδιαίτερα ατυχές δε, καθότι η διαβούλευση που έλαβε χώρα προκύπτει ότι έλαβε τις περισσότερες απαντήσεις που λάβαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα, ποτέ σε σχετική διαβούλευση. Επομένως, μια πληρέστερη διαβούλευση θα είχε λάβει ακόμα περισσότερες απαντήσεις και θα είχαμε ακόμα περισσότερη υποστήριξη, δικαιολόγηση για την κοινή γνώμη. Θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν ακολούθησε τη διαθεσμική συμφωνία στην περίπτωση αυτή. Και τέλος θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία του να υιοθετηθεί η οδηγία αυτή το συντομότερο δυνατόν, ιδανικά πριν το τέλος της παρούσας θητείας, το οποίο θα επέτρεπε στα κάτι μέλη να είναι σωστά προετοιμασμένα εν ώψη των νέων διατάξεων. Η Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού σχεδιάζει να έχει ψηφοφορία 4 Μαρτίου και να ξεκινήσει διαπραγματεύσει ώστε να μπορέσει να υιοθετηθεί στην Ολομέλεια Μάρτιο ή Απρίλιο. Η Γιούρη θα ψηφίσει στις 19 Φεβρουαρίου την επόμενη συνάντησή μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη που θα ήθελαν να σχολιάσουν. Επιτρέψτε μου πριν από αυτό να πω ότι τη Δευτέρα η Επιτροπή Τραν είχε εργαστήριο επί θέματος αυτού με το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε και το 2015 δηλαδή σημειώνονταν υπογραμμίζονταν προβλήματα για τη δημόσια υγεία. τις σχετικές πληροφορίες για τις μελέτες που έχουμε για τον αντίκτυπο στη δημόσια υγεία μπορείτε να τις έχετε επικοινωνώντας και με το προσωπικό μου γραφείο. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, το, για το σχέδιο αυτό. Καταρχάς ε, δύο βασικοί λόγοι που νομίζω ότι αποξάλλονται και από τη συζήτηση. Ο πρώτος είναι η επιπτώση στην υγεία ιδίω ό,τι αφορά ευαίσθητε επαγγελματικέ ομάδε ε, και κυρίω βέβαια ηλικιωμένου και μικρά παιδιά. Και επειδή και εγώ προέρχομαι από ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο που ζει τις αρνητικές επιπτώσεις ε, στη Γεωργία, είναι ένα παράδειγμα και αυτό αλλά σε ό,τι αφορά τις αλλαγές της ώρας ε, για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες υπάρχουν ε, πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Ε, τη Δευτέρα νομίζω ξεκαθαρίστηκε ότι υπάρχουν και επιχειρήματα για την οδική ασφάλεια που δεν ε, συνηγορούν υπερικατά της κατάργησης της αλλαγής της ώρας ε, και ό,τι αφορά τα οικονομικά επίσης. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στα οικονομικά επιχειρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ε, δεν έχει κάνει κάποια ε, πλήρη μελέτη αντικτύπου, οπότε αν λάβουμε υπόψη και την, ε, τον περιορισμό ε, διάρκειας της διαβούλευσης, θα πρέπει τώρα να λάβουμε μια απόφαση έτσι πολύ βεβαιασμένα και λυπούμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ως νομοθέτες ε, έχουμε την ε, ανάγκη να λάβουμε υπόψη την άποψη των 4,6 εκατομμύρων Ευρωπαίων που συμμετείχαν ε, στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες για την κατάρριξη της αλλαγής ώρας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια ομογενή ζώνη ώρας παντού. Αυτό, λοιπόν, το πρόβλημα παραμένει και είπατε για το 2021 να είναι τελευταία αλλαγή ώρας, να αναβληθεί δηλαδή ε, η ημερομηνία. Ε, ίσως αυτό θα βοηθήσει να βρεθεί μια λύση από τα κράτη-μέλη, ώστε να μην έχουμε μια μεγενή τέτοια αζώνη ώρας για Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάουφμαν. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. μάλλον να, να μην μακρηγορήσω, ε, δεν μπόρεσα να διαβάσω αναλυτικά την έκθεση, αυτή την παρουσίαση μάλλον, αλλά εκεί γίνεται λόγος για προβλήματα υγείας και δεν ε, το πιστεύω και πολύ αυτό, γιατί είναι τόσο δραματικά τα πράγματα τότε δεν θα έπρεπε να πηγαίνει κανείς διακοπές παίρνοντας και τα παιδιά του μαζί ή τους ηλικιωμένου ε, σε μια άλλη χώρα που έχει μεγάλη διαφορά ώρας. Αν ήταν τόσο δραματικές οι επιπτώσεις ε, ε, δεν θα πήγαινε κανείς να περάσει δύο εβδομάδες σε μια άλλη ζώνη ώρας στις διακοπές του γιατί είναι επιβλαβές αυτό για την υγεία του. Και τι κάνουν οι εργαζόμενοι σε βάρδιες τελικά. Άνθρωποι οποίοι όλη τους τη ζωή, δουλεύουν με νυχτερινή βάρδια τη μια εβδομάδα, ημερήσια βάρδια την άλλη εβδομάδα ε, και αυτό δεν το αναφέρουμε, αλλά εδώ το αναφέρουμε ε, ε, για την αλλαγή ως επιχείρημα την αλλαγή της μιας ώρας και πραγματικά νομίζω ότι τα υπερδραματοποιούμε τα πράγματα. Βέβαια όλοι ε, είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης και για τη Γερμανία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι είναι υπέρ της κατάρρησης αλλαγής ώρας. Αν συζητήσω σήμερα με Γερμανούς ε, συμπολίτες μου μπορεί να μου πούνε ότι ναι, δεν θα ήταν κακό να καταργηθεί αλλαγή ώρα, αυτό θα μου λέγανε. Όμως... Ε, ε, δεν θέλω ε, να μην... Ε, τι θα γίνει με τις αλλαγές, μάλλον τις διαφορετικές ζώνες ώρας, τις παραλλαγές αυτές που έχουμε, τις διάφορες εκδοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω κατά πόσο να οι Γερμανοί συμφωνούν ακριβώς ε, με τις ε, αλλαγές αυτές ε, που προτείνεται, δηλαδή κάποιοι να είναι στην θερινή, κάποιοι να είναι στη χειμερινή, πρέπει να βρεθεί μια συντονισμένη λύση ενδεχομένως. Πάντως δεν με έχει πείσει το επιχείρημα της υγείας. Κύριε Χάουταλ, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά αυτά που μας είπε μόλις η συνάδελφος η κυρία Κάουφμαν να πω ότι είμαι πεπισμένη ότι εδώ υπάρχει ένας παράγοντας που αφορά στην υγεία και η έκκληση πολλών συμπολιτών μας ε, να κάνουμε κάτι γι' αυτό δείχνει ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ε, τον ε, το ιστορικό μας ρολόι. Ακόμα και το γεγονός ότι κάθε μία ή δύο εβδομάδες αλλάζω το ωράριό μου κατά μία ώρα, αυτό με επηρεάζει. Ε, κοιμάμαι πιο αργά στο Ελσίνγκη, πιο νωρίς στις Βρυξέλλες, ε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Υπάρχει ένα δύσκολο ζήτημα εδώ για τις, τόσο για την υγεία για τους ε, εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν βάρδιες. Ε, είναι μεγάλος αντίκτυπος ε, για αυτούς που δουλεύουν ιδιαίτερα όταν είναι βάρδιες 8 ώρα και που αλλάζουν τη βάρδια τους συνεχώς και ποτέ δεν μπορούν να βρουν την ησυχία τους κατά κάποιο τρόπο. Ε, σχετίζεται δηλαδή και με την εργασιακή νομοθεσία τελικά. Θα έπρεπε να εκκριζωθούν οι χειρότερες μορφές ε, διατάραξης ε, της, του ύπνου των ανθρώπων, του, του βιολογικού ρολογιού και του, του, του σωματικού ρολογιού. Τώρα υπάρχουν και κάποιες πτυχές που έχουν να κάνουν με, τη, με τα νομικά. Πρώτα απ' όλα, αν για μια φορά μπορούμε να πάρουμε μια ορθολογική απόφαση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο καλά. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη σύγκληση μεταξύ κρατών μελών. Εμεί ω Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τις συζητήσει μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι ώστε, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, να φτάσουμε να κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια. Τώρα έχουμε αυτή την αιτιολογημένη γνώμη ε, του ε, Δανικού Κοινοβουλίου που αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Από τις 3 του Δεκέμβρη το έχουμε αυτό. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν ή ενδεχομένω κάποιο άλλο. Ε, τι πιστεύει για αυτό το ζήτημα της αρχής της επικουρικότητας. Εγώ δεν νομίζω να είναι θέμα επικουρικότητας. Μια και η εναρμόνιση έχει εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλουμε αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο στην ιστορική αγορά. Έτσι ξεκίνησε. Οπότε δεν βλέπω πώ εδώ μπαίνει θέμα επικουρικότητα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτή η γνώμη. Τέλο, να πω ότι ναι, χρειάζεται αυτή η καθυστέρηση, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα κράτη-μέλη δεν προσπαθούν πια να βρουν λύση και τελικά τελευταία στιγμή να υπάρξει μια κρίση πρώτου αδιεξόδου. Είναι όπως το Brexit αν θέλετε, ε, σε άλλη κλίμακα βέβαια. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί πάντως πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετόν έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ είμαι υπέρ τη κατάργηση αυτή τη αλλαγή τη ώρα. Χαίρομαι που επανέρχεται εδώ αυτό ο φάκελο. Θυμάμαι ότι είχαμε συζητήσει ήδη το 2015. Τότε απέτυχε αυτό το εγχείρημα, αλλά σίγουρα δεν έφταιγε γι' αυτό η Επιτροπή μα. Είναι πολύ καλό που επανέρχεται το ζήτημα. Όπω ελέγχθη, υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κατάργηση αυτή. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα θέμα δημόσια υγεία, μια και η αλλαγή ώρα ε, διαταράσει το βιολογικό ρολόι, δημιουργεί κούραση, δημιουργεί κίνδυνο για ατυχήματα. Ένας άλλος λόγος που δεν έχει, ο οποίος δεν έχει αναφερθεί είναι ότι θα ήταν κάτι θετικό για τη γεωργία, διότι η αλλαγή της ώρας ε, διαταράσει μεταξύ άλλων ε, και το άρμεγμα των αγελάδων, την, τον ρυθμό ζωής των ζώων και βεβαίως ο τρίτος λόγος και ο πιο σημαντικός είναι ότι είναι αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Μία και όλα τα στατιστικά, όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια συντριπτική πλειοψηφία Ευρωπαίων θέλουν να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας. Και η δημόσια διαβούλευση που έκανε η Κομισιόν το αποδεικνύει. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι ερωτήθηκαν και 84% εξ αυτών ε, είναι υπέρ της κατάργησης. Οπότε δεν νομίζω να πρέπει να διστάσουμε εδώ και δεν υπάρχει και κάποιο, κάποιο νομικό κόλλημα. Δεν ανησυχώ τόσο για το θέμα τη νομική βάσης. Τα έγγραφα που μα μοιράστηκαν το, το δείχνουν. Αυτό μπορούμε να ε, επικαλυστούμε το άρθρο 114 της συνθήκης για την σωστή λειτουργία τη αγοράς αγορά ε, για ένα τέτοιο μέτρο. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε αυτή την κατάργηση. Εγώ πάντα την υποστήριζα και πριν γίνω Ευρωβουλευτής. Είμαι μεταξύ αυτών των 84% των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λοτόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα σας ευχαριστήσω ε, για την παρουσίαση αυτού του σχεδίου, αυτού του draft. Ε, χθες ε, συμφωνήσαμε αλλά σήμερα με τον κύριο Βόλκαν, αλλά τώρα δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι κατοπαροκέ αγελάδε. Ε, ε, θα κατεβάσω περισσότερο γάλα άμα να καταργηθεί η αλλαγή ώρα. Κατά πάσα πιθανότητα κάπως προσαρμόζεται ο οργανισμός ε, από μόνος του σε αυτές τις αλλαγές. Δεν ξέρουμε. Οι ειδικοί που μιλάνε για επιπτώσει στο τομέα τη υγεία, ε, ούτε και εμένα με πείθουν ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι η αλλαγή ώρα ε, υποτίθεται ότι είχε γίνει για την εξοικονόμηση ενέργεια, αλλά τώρα αυτό δεν ισχύει πια. Δηλαδή δεν εξοικονομείται πλέον ενέργεια με την αλλαγή ώρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε ό,τι την κατάργηση τη αλλαγή ώρα, ε, σίγουρα χρειάζεται και τη στήριξη από πλευρά κοινή γνώμη. Πολλοί όμω αμφιβάλλουν πώ ακριβώ θα γίνει αυτό. Και σε ό,τι αφορά τι αιτιολογήσει και τα επιχειρήματα, τέλο πάντων, θα πρέπει να δούμε. Ε, τώρα, έρχομαι σε κάποια στοιχεία μεμονωμένα. Στην πρόταση Κομισιόν. Αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν δεν μας φαίνονται ρεαλιστικά. Και το είδαμε και στην Επιτροπή Μεταφορών. Και νομίζω ότι τα δύο χρόνια είναι μια ελάχιστη προθεσμία για την οριστική μετακατάργηση της αλλαγής ώρας. Τώρα το να μιλάμε για ε, προθεσμίες σταθερές, ε, το θέμα είναι πότε θα το αποφασίσουμε. Για νομίζω ότι χρειάζεται ευελιξία. Και όχι να πούμε τώρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω πίσω ότι έχει τεκμηρώσει επαρκώ την πρότασή σα. Εδώ θα συμφωνήσω με τον ε, κύριο Βέλκεν. Επομένω. Και για τα κράτη-μέλη. Ναι, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτό ε, θα πρέπει να αναφέρεται και στην ε, σχετική οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε, Ελπίζω να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης να επηρεάσει, να το απολογή σε αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ. κυρία Χανιμπολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Χαούταλα. Και οι δύο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αλλάζουμε ώρα κάθε εβδομάδα, λέει ο Μιλήτρια. Και είναι κουραστικό είναι επιβαρυντικό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν με πείθει το πρόβλημα δημόσιας υγείας για, τις, ε, για την αλλαγή διαφορές στον χρόνο. Εμείς έχουμε επιβιώσει ταξιδεύοντας ακόμα και αν είναι κουραστικό. Νομίζω ότι τα προβλήματα υγείας είναι ένα αμφίβολο θέμα. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα βοηθούσε στο συντονισμό. Η αλλαγή της ώρας γίνεται από όλους την ίδια στιγμή. Δεν αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία συντονισμού. Εφόσον γίνεται η αλλαγή η εποχιακή της ώρας την ίδια στιγμή, εγώ ήμουν στην Επιτροπή Μεταφορών το 2000 και ασχολούμαι με το θέμα, με ενδιαφέρει εδώ και αρκετό καιρό. Πάντως πρέπει να πω ότι η διαβούλευση δεν ήταν τόσο ευρεία όσο θα μπορούσε να είναι. Γνωρίζω ότι τα 4,5 εκατομμύρια είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, αλλά συνολικά στο σύνολο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρός αριθμός και αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα μου άρεσε να είχαμε μια διαβούλευση πορίσματα πολύ ευρύτερης μελέτη διαβούλευσης. Και βεβαίως εδώ μιλούμε κυρίως για τις αλλαγές από Ανατολή προς Δύση, αλλά υπάρχουν και οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τελείως διαφορετικές οι περίοδοι φωτός από τα βόρεια της χώρας μέχρι τα νότια. και ίσως ε, η αλλαγή της ώρας βοηθάει για το μισό της χώρας να έχει περισσότερο φως. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και σε άλλα κράτη-μέλη, αν είναι θέμα ή όχι, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και το γεωγραφικό πλάτος και όχι μόνο το μήκος. Επομένως υπάρχουν πολλές τυχές. μαζί με την περιορισμένη διαβούλευση θεωρώ ότι το πράγμα έχει προωθηθεί υπερβολικά ταχαίως. Η δε μεταβατική περίοδος η δεν μας φαίνεται και τόσο μακρά. Μιλούμε για εποχιακή αλλαγή που σημαίνει δύο φορές το χρόνο και μέλος μιλούμε για τέσσερις αλλαγές συνολικά. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στα πλαίσια αυτής εδώ της Επιτροπής. Φαίνεται όμως ότι έχει προωθηθεί λίγο βιαστικά το θέμα και δεν είμαι βέβαιη ότι έχουμε σκεφτεί το σύνολο του αντικτύπου. Σας ευχαριστώ η Γκέριγκερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, ο λόγος της υποβολής, ε, μάλλον της εισαγωγής της εποχιακής έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχει πια πλεονέκτημα δηλαδή που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από την εποχιακή αλλαγή ώρας και επομένως γιατί να τη διατηρήσουμε. Δεν ενέχει πλεονεκτήματα και απλώς περιπλέκει τη ζωή μας. Και εδώ το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να κινείται υπερβολικά γρήγορα Δηλαδή όλοι ελπίζουν ότι το Μάρτιο θα αλλάξουν, μάλλον έχουν όλοι προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι το Μάρτιο θα αλλάξουν για τελευταία φορά την ώρα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να έχουμε πολύ μακροσκελής ε, περιόδους ε, μεταβατικές. Δεν είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε, να αλλάζουμε τους ε, δείκτες του ρολογιού. και νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει υπερβολικά. Γνωρίζουμε ποια είναι η επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών και δεν πρέπει να εμένουμε στην αντίρρηση προς αυτή την επιθυμία. Και σας βεβαιώ ότι δεν είναι ότι θα έχουμε περισσότερο ή λιγότερο ηλιακό φως. Το ηλιακό φως είναι αυτό που είναι ακριβώς τόσο. Δεν χρειάζεται καμία μετάβαση. Απλώς κάποια ορισμένη στιγμή δεν θα ξαναλλάξουμε την ε, ώρα και θα συνεχιστεί η ζωή μας όπως ήταν. Θεωρώ ότι είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές γιατί έτσι οι πολίτες θα δουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές. Ε, έχουμε παίξω που αναμένουν και ε, θα ήθελα να ακούσουμε πολύ σύντομα παρακαλώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε τα μέλη και ε, τον εισηγητή. Να ευχαριστήσουμε για τα θετικά σχόλια που έχουν γίνει σχετικά με την πρόταση αυτή. Σημειώνουμε ότι διατηρείται την ανάγκη μιας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών και εναρμονισμένης προσέγγισης και για το μέλλον για τις εποχιακές αλλαγές της ώρας. Σημειώνουμε επίσης τα σχόλια που έγιναν σχετικά με τον χρόνο, την περίοδο μετεγραφής και την περίοδο υλοποίησης. Έχουμε πράγματι τοποθετήσει, υποβάλει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα με την υπόθεση εργασίας ότι οι συνομοθέτες θα συμφωνούσαν προτού ολοκληρωθεί η παρούσα θητεία του Κοινοβουλίου. Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, ε, θα εξαρτηθεί, εν πάση περιπτώσει, από τους συνομοθέτες η τελική απόφαση. Για ένα σχόλιο που έγινε σχετικά με την επικουρικότητα, να σας ενημερώσω ότι είχαμε μία συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Συμβούλιο. Η νομική υπηρεσία της Κομισιόν έχει γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου απήντησε στο σχετικό ερώτημα, συμφωνώντας με την πρόταση της Κομισιόν, χωρίς να βλέπει δηλαδή κάποια απόκληση από την αρχή της επικουρικότητας και σχετικά με την χρηστή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς για τις αρχές ε, της χρησιμοποίησης των αξιολογήσεων αντικτύπου πράγματι προχωρήσαμε σε μια δημόσια διαβούλευση που ήταν βραχύτερη από την κανονική της διάρκεια που είναι 12 εβδομάδες. Παρόλα αυτά σπάσαμε όπως υπόθηκε κάθε ρεκόρ από τον αριθμό των απαντήσεων. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να υποβάλουμε, να είμαστε έτοιμοι να έχουμε χρόνο ή στην παρούσα θητεία του Κοινοβουλίου να συζητηθεί το θέμα και να φτάσουμε σε μια απόφαση. Αυτό εξηγεί το χρονοδιάγραμμα υποβολή τη προτάσεω μας. Αλλά θυμίζουμε ότι δεν πρόκειται για μια καινούργια θεματική, είναι κάτι που έχει επανέλθει διάφορες φορές τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που έχουμε παρακολουθήσει στενά στην Κομισιόν. Διαβάζοντας το επεξηγηματικό μνημόνιο θα δείτε όλες τις ενδείξεις που έχουμε συλλέξει και την ίδια τη μελέτη του 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρούμε απόλυτος επικαιροποιημένη που περιγράφει αναλυτικά όλες τις πτυχές του αντικτύπου. Και η τελευταία ομιλήτρια είπε ότι αυτό ήταν πίσω από τους αρχικούς λόγους της υποβλήσης Κομισιόν, δηλαδή η ενεργειακή εξοικονόμηση, οι ενδείξεις που έχουμε ε, μας λένε ότι η οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενεργειακή είναι περιθωριακή. Για την, δηλαδή, της εποχιακής αλλαγής της ώρας. Έχουμε συγκεντρώσει όλες τα, τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαμε επί των μεταφορών, επί των ε, μετακινήσεων εργαζομένων, της δημόσιας υγείας. Υπάρχει βεβαίως ένα κόστος αλλαγής των συστημάτων, αλλά θα ήταν ad hoc. Ε, με μεταβατική περίοδο δεν θα είχαμε πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά θα είχαμε πρόσθετο όφελος για τους πολίτες, οι οποίοι δεν θα είχαν πλέον απορία για το πότε αλλάζει η ώρα, δηλαδή κάθε έξι μήνες. Ευχαριστώ. All the ε, Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Βεβαίως είναι πάντα ένας πειρασμός να συζητούμε αυτό το θέμα, όμως ε, τα ζητήματα υγείας δεν είναι δική μας αρμοδιότητας. Μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στην ακρόαση του 2015 καθώς και στο εργαστήριο εχθές για να πειθούμε γι' αυτό η συντονισμένη προσέγγιση τους ή άλλως ε, είναι κάτι το οποίο είναι κόκκινη γραμμή για όλους. Εδώ δεν πρέπει να το φοβόμαστε αυτό και να έχουμε κατά νου ότι το πέρασμα από τη χειμερινή στην καλοκαιρινή ώρα, στη θερινή ώρα, δεν είναι ότι η μέρα γίνεται 25 ώρες, έτσι. 24 είναι οι ώρες. Δεν προσποιούμαστε ότι το καλοκαίρι έχουμε 25 ώρες ξαφνικά. Η κυρία Κάουφμαν αναφέρθηκε στις δύο ωριές άτρακτους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι θα έχουμε μία. Τώρα το θέμα που έθεσε η Δανία, ε, το θέμα αρμοδιότητας δηλαδή, πριν από λίγες μέρες μίλησα με τον Τσέχο Υπουργό που είπε ότι θεωρεί ότι αυτός ο τομέας ε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντελώς αντίθετη θέση δηλαδή από αυτή της Δανία. Το λέω για να το προσθέσω και αυτό στη συζήτηση. Θα είχα να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους λόγους για τους οποίους η νομοθετική πρόταση υπευλήθη τώρα, Μια συντομία όμως γιατί έχω και μια, μια επιστολή από το 2016 από την Επίτροπο Μπουλς που λέει ότι δεν θα εξετάσει το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι κάτι δευτερεύον. Μπορεί να άλλαξε έκτοτε από η μετά τη δημόσια διαβούλευση βέβαια. Λοιπόν, κλείνουμε με το θέμα αυτό και θα καλέσω το προσκεκλημένο μας τον ε, Ρουμάνο Υπουργό τον κύριο Τοάντερ να έρθει στη συνάντησή μας.

So, dear colleagues, I Αξιόριμοι συνάδελφοι, καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Τουντορέλ Τοάντερ, που εκπροσωπεί τη Ρουμανική Προεδρία που θα μας παρουσιάσει, και θα μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη Ρουμανική Προεδρία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου. Συμπίπτει βέβαια αυτή η περίοδος με το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου. Είναι μια φορτωμένη περίοδος για, τις δύο, για τα δύο θεσμικά όργανα. Αναμένω να ακούσω τι προτεραιότητε ε, της Προεδρία στον τομέα, στους τομείς που ε, μας απασχολούν. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω στον Υπουργό. Θα πρότεινα να του δώσουμε 20 λεπτά το λόγο και στη συνέχεια θα έχουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας, όμως στα δύο χρόνια που είμαι υπουργό δικαιοσύνη, έχω συναντήσει κάποιους από εσά. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα και είμαι περήφανος που θα παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανίας και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Έχω ετοιμάσει κάποιες μικρές αναφορές για όλους τους φακέλους που αφορούν τη δικαιοσύνη και που έχουμε ε, κληρονομήσει από την ε, Αυστριακή Προεδρία, αλλά θα αναφερθώ όλους ιδιαίτερως ε, στα ζητήματα από τον οποίων εργαζόμαστε τώρα και βεβαίως τους φακέλους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής σας. Ως υπουργό Δικαιοσύνης, πρώτα απ' όλα θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σύνολό του, Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι δραστηριότητές σας, το έργο σας εδώ, με βάση πάντα βεβαίως τις αρμοδιότητες που έχει κάθε επιτροπή, είναι το υψηλότερο επίπεδο έκφρασης το ιδεώδους της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Αυστριακή Προεδρία από την οποία πήραμε τη σκητάλη και με την οποία είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία κατά την προπαρασκευή της Προεδρίας μας. Από κοινού με τους συναδέλφους τους είμαι επίσης εξαιρετικά ευγνώμων είτε προέρχονται ε, από την μόνιμη προσωπία είτε από το Υπουργείο ε, μπορέσαμε σιγά σιγά να εξοικειωθούμε με τους διάφορους φακέλους ε, που θα μας απασχολούσαν, την εξέλιξή τους, έτσι ώστε όταν πια αναλάβαμε την Προεδρία, γνωρίζαμε το περιεχόμενο αυτών των ε, φακέλων, τα καλά τους, τα κακά τους, τι ακριβώς έμενε να κάνουμε, Έτσι λοιπόν, με βάση τα που έχουν επιτευχθεί, προσπαθούμε να προωθήσουμε τους φακέλους αυτούς έτσι ώστε να μεταφραστούν σε νόμους. Και βεβαίως ε, θα σεβαστούμε όλους τους κανόνες, όλα όσα πρέπει και μπορεί να κάνει μια Προεδρία του Συμβουλίου. Δεν ε, θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση για τα πάντα. Δεν είμαστε ε, αγαθοί. Μπορούμε όμως να τα βρούμε για κάποια ζητήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μία συνένεση, συμβιβασμού έτσι ώστε η νομοθετική διαδικασία να προχωρήσει όσο γίνεται περισσότερο. Προσωπικά, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές ρυθμίσεις υψηλού επίπεδου έτσι ώστε τα ωφέλη από αυτές τις πολιτικές και από αυτά τα πρότυπα τελικά που προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτήν την διαδικασία νομοθεσίας και θέσει προτύπων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία δεν έχει επιστροφή. Οι ωφελημένοι λοιπόν να είναι οι πολίτε αυτή τη διαδικασία. Διότι οι πολίτε είναι αυτοί που ελπίζουμε θα εμπιστευτούν στη συνέχεια αυτές τις διαδικασίες είναι αυτοί που θα υποφεληθούν αυτού του καταπληκτικού και γενναιόδωρου σχέδιου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησα σήμερα και στην Επιτροπή Ελευθεριών και μία ευρωβουλευτής ε, είπε ότι η Ρουμανία πρέπει να είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Και το εκτίμησα αυτό που είπε αυτή η ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω αν η Ρουμανία είναι όντως στην καρδιά της Ευρώπης, Διότι είναι δύσκολο να πει κάνεις. Ε, ποιο είναι στην καρδιά τη Ευρώπη. Η καρδιά είναι ούτω ή άλλω ένα περίπλοκο όργανο. Αυτό που μπορώ να σα πω όμω σίγουρα είναι ότι η Ευρώπη είναι στην καρδιά, είναι στις καρδιές των Ρουμάνων. Οι στατιστικές, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Ρουμάνοι είναι από τους πιο φιλοευρωπαίους, ε, είναι από τους πιο πεπισμένους για τα ωφέλη ε, της Ευρωπαϊκής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της. Ξέρετε, περάσαμε από κομμουνιστικό καθεστώς και πάντα η Ευρώπη ήταν για μας ε, ένα χώρος ασφάλειας, ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε τις ελευθερίες που μας λείπουν, έναν χώρο όπου μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας και όπου μπορούμε να πετύχουμε ε, τους στόχους μας, τις προσδοκίες μας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου ελπίζει να έχει μια στενή, καλή, επικοδομητική συνεργασία με με την Επιτροπή σας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τους άλλους συνομοθέτες. τα πλαίσια πάντα και με βάση τα όρια των αρμοδιοτήτων του καθένα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και πρέπει όλοι να σεβόμαστε. Τώρα θα περάσω σε ορισμένα πιο συγκεκριμένα πράγματα, αλλά να κάνω ακόμα ένα γενικό σχόλιο. Οι αρχές βάσει των οποίων θα ασκήσουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων είναι γενικές αρχές. Μπορούν όμως επίσης να, να μεταβληθούν σε συγκεκριμένα βήματα με βάση τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Σεβασμός των κοινών αξιών, σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και βεβαίως σεβασμός του κράτους δικαίου. Σεβασμός ε, των διαφόρων συστημάτων και παραδόσεων και στον τομέα του δικαίου, οικοδόμηση αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο αναλάβουμε εμείς την Προεδρία και θα την ασκήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας. και στον τομέα της δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Εγώ ειδικεύομαι σε αυτόν τον τομέα και πάντα εκτιμούσα τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζετε εσεί ε, στη διαδικασία ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ελπίζουμε μαζί με εσά να μπορέσουμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το έργο, το νομοθετικό, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει όλοι μας ως μέλη της Ένωσης αλλά και ο καθένας προσωπικά όσοι εργάζονται σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Θέλουμε να ενσωματωθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ήρθα λοιπόν εδώ σήμερα με βάση την ιδιότητά μου αυτή και ήρθα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Ήρθα εδώ με τους 15 νομοθετικούς και μη νομοθετικούς φακέλους που κληρονομήσαμε από την Αυστριακή Προεδρία και σε ένα περισμένο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να αναφερθώ στους φακέλους εκείνους όλος ιδιαίτερος όπου συμμετέχετε κι εσείς και όπου έχετε αποφασιστικό ρόλο. Για τη Ρουμανική Προεδρία, μια προτεραιότητα είναι ο κανονισμός του Συμβουλίου για την ε, δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε ζητήματα χαμικού ε, δικαίου, ε, Γονική ευθύνη ε, και απαγωγή παιδιών. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά βέβαια. Δεν θα πω σε λεπτομέρειε, αλλά θα αναφερθώ σε κάποιες ιδιαιτερότητε. Στη Ρουμανία, εμείς ε, πλέον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Η νομοθεσία αυτή λοιπόν είναι απαραίτητη, διότι θα έρθει να διευκρινίσει, και πρέπει να συμβεί αυτό, κάποιες καταστάσεις και στην πραγματικότητα αλλά και νομικά καταστάσεις που δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια. Και εμείς θα κάνουμε κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της, ομα, ε, αλλά και στο Συμβούλιο επί τη βάση της γενικής προσέγγισης ότι το Συμβούλιο Τζάι, ε, που μάλλον στην οποία έφτασε το Συμβούλιο Τζάι το Δεκέμβριο, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία έως το τέλος ε, της θητείας μας. Έως δηλαδή τα τέλη Ιουνίου 2019. Το οικογενειακό δίκαιο και ε, το συμφέρον του παιδιού αποτελούν προτεραιότητα, για μας και η γνωμοδότησή σας του Ιανουαρίου του, του 2019 είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας διότι εμείς συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο και συμμεριζόμαστε και τις ίδιες αξίες. Ως το επιχειρησιακό σκέλος της, ε, ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2α που έχει συμφωνηθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2018 η Ρουμανική Προεδρία θα ολοκληρώσει το προήμιο και θα αρχίσει να εξετάζει μέρος του εγγράφου και θα προετοιμάσουμε κάποιες διατάξεις ε, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι πρέπει να ακουστεί η άποψη του παιδιού. Η οδηγία για όσους ε, ε μεταφέρουν παρατυπίες και παραβίαση νομοθεσίας ενωσιακής, τους λεγόμενους whistleblowers, αποτελεί προτεραιότητα για μας. Το λέω αυτό, βεβαίως θα μιλήσω και θα πράξω ως πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία από τον τομέα αυτόν. Βεβαίως μπορούμε να βελτιώσουμε και τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους whistleblowers. Γιατί το λέω αυτό. διότι από το 2004 υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μου για τους whistleblowers και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες whistleblowers διαφορετικές κατηγορίες, διάφορες βαθμίδες αν θέλετε σε ό,τι αφορά τι κυρώσει που μπορούν να υποστούν από τις αρμόδιες αρχές. Για μας λοιπόν αυτό αποτελεί προτεραιότητα και έχουμε έτσι μεγάλες προσδοκίες να ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο. Η πρόοδος που σημειώθηκε επί αυστριακή Προεδρίας είναι κάτι θετικό. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο και ελπίζουμε να επιληφθεί αυτός ο στόχος τομέα των δυνατόν. Η αλλαγή του κανονισμού του Συμβουλίου για τα πολιτικά στοιχεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη ανάγνωση, η τροποποίηση του σχετικού κειμένου. Όμως ε, θα πρέπει ε, να δώσουμε συνέχεια στον φάκελο αυτόν στην κατάσταση στην οποία το βρήκαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό. Και βεβαίως ε, όλες οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών χρειάζονται αυτό το μέσο, χρειάζονται αυτό το σύγχρονο εύκολο τρόπο να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για μια πιο γρήγορη και πιο εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται ούτε εδώ να μπω στην ουσία του φακέλου, μιας και σχετίζεται με την αποστολή ετοιμάτων ε, για αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια. Εδώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη εξυγχρονισμού της δικαστικής συνεργασίας σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Για να κάνω μια σύγκριση, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, στην Επιτροπή Ελευθεριών, μίλησα για ηλεκτρονικά ε, στοιχεία σε ποινικέ υποθέσεις σε ό,τι αφορά την αποθήκευση αυτών των στοιχείων με τον ορισμό ενός εθνικού εκπροσώπου που παρακολουθεί όλα τα αιτήματα από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα όμως να κάνω μία σύγκριση. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί. Εάν δούμε την εκπόνηση μιας νομοθεσίας ε, για ζητήματα δικαιοσύνης ε, σε ποινικό επίπεδο και εκεί μιλάμε για την χρήση μοντέρνας τεχνολογίας ε, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά στοιχεία και σε αστικά και εμπορικά ζητήματα. <coughs> Εμείς καλωσορίζουμε το γεγονός ότι εγκρίνατε την έκθεση της, του κυρίου Ράντεφ και εμείς εκφράσαμε, εκφράζουμε την ελπίδα μας ότι οι εμπειρογνώμονες, οι συνάδελφοι, σε συνεργασία μαζί σας, θα μπορέσουν να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτού του φακέλου. Τώρα, ο κανονισμός για την επίδοση εγγράφων. Και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής σας τον Δεκέμβριο 2018. Αυτή η πρόταση έρχεται να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, ζητήματα αστικού δικαίου. Όλοι θέλουμε μια πιο αποτελεσματική και μια πιο φτηνή δικαιοσύνη για τους συμπολίτε μας, για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε τα δικαιώματα των ε, εμπλεκομένων να διαφυλαχθούν καλύτερα. Μιλάμε εδώ για αστικό δίκαιο, μιλάμε για δικαιωμα... Ε, διαδικαστικά δικαιώματα. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση εδώ για ποινικό δίκαιο. Η υποχρέωση που έχουν τα δικαστήρια να έχουν ηλεκτρονικά έγγραφα θα έρθει να αλλάξει όλες τις προδιαγραφές αλλά και όλες ε, τις διαδικασίες στις διάφορες χώρες και η Ρουμανική Προεδρία θα καλέσει το Συμβούλιο να φτάσει σε γενική προσέγγιση για το θέμα αυτό στη συνάντηση 6 και 7, που θα γίνει 6 και 7 Ιουλίου του 2019. Ο κανονισμός τώρα που έχει να κάνει με τις προσφυγές, την καταγραφή των προσφυγών, αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου για τις κεφαλαιαγορές, Θέλουμε να αυξηθεί η διασυνοριακή εξέταση προσφυγών θέλουμε εδώ να αυξηθεί η νομική ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά. Το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα ζητήματα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος θα, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε τρίτους στις περιπτώσεις αυτές και να βρεθεί το κατάλληλο πεδίο που θα καλύπτει αυτός ο κανονισμός. Ε, εμείς καλούμε την Κομισιόν να συμφωνήσουν, να συμφωνήσει ε, σε μια συζήτηση προσανατολισμού ή να φτάσουμε σε γενική προσέγγιση, προς περιπτώσεις μέσα από μια συζήτηση στην συνάντηση αυτή στις 6 και 7 Ιουνίου του 2019. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο που έχει να κάνει με το εταιρικό δίκαιο που περνάει από τη σύνθεση διαδικασία ε, σκοπεύουμε, ελπίζουμε να υπάρξει σύμφωνη γνώμη από το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόταση για την ψηφιοποίηση διότι εδώ το Συμβούλιο ήδη έχει λάβει διαπραγματευτική εντολή. Η οδηγία τώρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και μετατροπές εδώ υπάρχουν κάποια τεχνη, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να επιληθούν πριν φτάσουμε σε συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου και έχει γίνει και μια συζήτηση η οποία όμως τελικά λύθηκε η παρεξήγηση που δημιουργηθεί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. είναι ένα θέμα που για μένα προσωπικά πέρα από την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Συμβουλίου ε, είναι ένα θέμα που, με, μου αρέσει ιδιαίτερα, που με ενδιαφέρει. Έχω μεγάλες προσδοκίες φάκελος φάκελο που εξετάζεται τώρα στην Επιτροπή Ελευθεριών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ορίσουμε ποιο θα είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέα, ποιο θα είναι, ποιος θα είναι ο Εθνικό Εισαγγελέα, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίω ε, χρειάζονται οι απαραίτητοι οικονομικοί αλλά και ανθρώπινοι πόροι για να αρχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία αυτή τα γραφεία, τα, ιέδρα, έδρα θα πρέπει να ε, αποφασιστεί το πού θα είναι ακριβώς. Ε, όλοι έχουν προσδοκίες. Να κάνω εδώ μια σύγκριση. Ε, εφόσον έχουμε Ευρωπαίους δικαστές, χρειαζόμαστε και Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εφόσον υπάρχει εγκληματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απάτη κατά του συμφερόντων της Ένωσης, εάν σε εθνικό επίπεδο ποινικοποιούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με απώλεια εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έχει μια διεθνή διάσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τους κατάλληλους θεσμούς που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουμε δημιουργήσει αυτόνομα, ε, ανεξάρτητα θεσμικά όργανα που θα προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι λαμβάνει η χώρα μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει η περίπτωση να διαβερνηθούν αυτές τις θερμοδιότητες και να συμπεριλάβουν και ζητήματα τρομοκρατίας, ε, νομιμοποίησης εσόδων, ε, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 86 συνθήκης. Δηλαδή, θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να έχουμε έναν Ευρωπαίο Εισαγγελέα, να έχουμε το κολέγιο των εισαγγελέων που θα εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη, να είναι όλα αυτά λειτουργικά, να επιχειρούν και μετά να συζητήσουμε για περαιτέρω αρμοδιότητες τροποποιώντας ενδεχομένως το άρθρο 86 της συνθήκης. Τώρα, το πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες. Εδώ μιλάμε για έναν τομέα που δεν είναι βέβαια τόσο αυστηρός όσο το ποινικό δίκαιο, αλλά δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο έτσι ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα έτσι ώστε να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών και όλοι οι πολίτες για την πραγματοποίηση όλων αυτών των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τους whistleblowers, παραδείγματος χάρη, και τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, κατά τη γνώμη μας, εμείς στο Βουκουρέστι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και σε νομικά ζητήματα. Δεν μιλάω εδώ τώρα για κάτι εξειδικευμένο, αλλά είναι σημαντικό ο Ευρωπαίος πολίτης να είναι κάπως εξοικειωμένος με τις βασικές νομικές αξίες της χώρας του, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, βλέπω ότι έχει περάσει ο χρόνος. Μίλησα λίγο περισσότερο από ότι μου αναλογούσε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε και σας ευχαριστώ κυρίως που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω εν συντομία τις προτεραιότητες μας Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν και κάποιες ερωτήσεις στις οποίες θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πραγματικά υπάρχουν ερωτήσεις ε, από τους ε, βουλευτές. Θα ακούσουμε όλους τους βουλευτές και εν συνεχεία θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε συνολικά. Κύριος Ντυρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού μου τυχε ο κλήρος να πάρω πρώτο το λόγο να καλωσορίσω τον Υπουργό, φυσικά. Σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Όπως και ο Πρόεδρος χαίρομαι και εγώ που άκουσα ότι είστε προσιλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μια από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος δικαίου. η τήρηση των κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη. Το λέω αυτό κύριε Υπουργέ, διότι φαντάζομαι έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει μία έντονη συζήτηση σε σχέση με τα τετάγματα που θέλετε να περάσετε στη δική σας χώρα. Αφού μιλήσατε για τη Ρουμανία, θέλω να σας πω ότι θα υπήρχε αμνίστευση πολλών προσωπικότητων, αν ψήφισαν αυτό το διάταγμα, και αυτό αντικείμενο έντονων συζητήσεων δεν είναι δε κατανοητό και από πολλούς νομικούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από επεσπιστές ε, του κράτους δικαίου. Σίγουρα δεν είναι εδώ ε, ο κατάλληλος χώρος για να έρθουμε σε παράθεση, Απλά σημειώνω το γεγονός ότι θέλετε να είστε ένα ενεργό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχετε μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις υπενθυμίζω. Δύο θέματα με ενδιαφέρουν περισσότερα. Δεν είναι εδώ κυρία Ρέγνερ που είναι η συγκήτρια για το εταιρικό δίκαιο, company law. Είπατε ότι θα προσπαθήσετε να λάβετε εντολή για να ολοκληρωθεί το θέμα πριν ε, το τέλος της δικής σας προεδρίας. Το δεύτερο θέμα είναι οι καταγγέλλοντες whistleblowers. Σε ευχαριστώ που είπατε ότι θέλετε να είναι προτεραιότητα της Προεδρίας σας αυτό το θέμα, όμως λίγο πιο συγκεκριμένα. Ποια είναι η θέση σας. Έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η θέση της Ρουμανίας απέναντι στην εξαίρεση της φορολογίας από το κείμενο. Ένα κείμενο πολύ σημαντικό για όλους μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Γκέριγκερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε εδώ και μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι σίγουρα κάτι σημαντικό. Και σίγουρα θα αποκτήσετε και πολλές εμπειρίες. Και ο στόχος είναι αυτός άλλος, να αποκτήσουμε όλη κοινή εμπειρία. Έχουμε και τις ευρωεκλογέ. Μέχρι τον Απρίλιο θα πρέπει λίγο πολύ να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας. Εσείς έχετε ένα εξάμεινο ε, ουσιαστικά, αλλά μειώνεται ε, ο φέλιμος χρόνος. Είναι κάπως ε, πετσοκομμένη, αν μπορώ να το πω έτσι, η προεδρία σας σε τέσσερις περίπου μήνες. Σίγουρα γνωρίζετε τις υποχρεώσεις ε, που υπέχετε και εσείς ε, και εμείς οι πολιτικοί και επίσης το πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης το γνωρίζετε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ένα παράδειγμα. Κατάργηση της αλλαγής ώρας. Είναι ένα θέμα. Το συζητήσαμε πριν από λίγο στην Επιτροπή μας. Το ερώτημα είναι αν είναι και αυτή προτεραιότητα για τη Ρουμανική Προεδρία, διότι αυτό είναι ένα αίτημα των πολιτών, όπως φάνηκε, η κατάρριξη δηλαδή. Και εν ώψη και των ευρωεκλογών σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι το Μάιο να έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Επίση, μεταρρύθμιση ό,τι αφορά τα δικαιώματα δημιουργού. Είναι ένα θέμα που το επεξεργαζόμαστε εδώ και τρία χρόνια. Είμαστε λίγο πριν ε, το σημείο τερματισμού, αν θέλετε. Έγιναν κάποιοι τερμερείς διάλογοι ε, και ελπίζαμε να υπάρξει ε, λύση του, και λήξη του θέματος, αλλά δυστυχώς υπήρξε εμπλοκή προσφάτως. Πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε να λυθεί το αδιέξοδο ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι με πολλές προεδρίες έχουμε συνεργαστεί για το θέμα αυτό και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να κλείσει. Γιατί ε, θα πιστωθεί στι επιτυχίες σας ε, ως Ρωμανική Προεδρία αν καταφέρετε να ολοκληρώσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Je vous remercie, je me joins. Κύριε σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σκεπτόμενος στη χώρα σας, σκέπτομαι ένα έθνος, ένα λαό που έχει υποφέρει πολύ με μεγάλα πλεονεκτήματα και μεγάλα ίσως μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ο πατέρας Μοσκοβισή, ψυχαναλυτής, που εγκατέλειψε τη χώρα του και που ήρθε στη Γαλλία, όπως πάρα πολλοί άλλοι συμπατριώτες του, ο Ντίνου Λιπάτη, μεγάλος πιανίστας, που είχα την τύχη να γνωρίσω, αλλά σκέπτομαι και δυσάρεστες πτυχές, <clears throat> πολιτικά συστήματα που υπό τα οποία υπέφερε η χώρα σας και μεγάλα κομμάτια της Ευρώπης. Άνθρωποι οι οποίοι κατέδωσαν την οικογένειές τους, ε, τις οικογένειές τους για να ανέλθουν ε, υπό το καθεστώς Τσαουσέσκου. Και σήμερα λοιπόν που η Ρουμανία η χώρα σας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σας ε, <clears throat> ζητούσα, θα σας ενθάρρυνα μάλιστα να μην προσεγγίσετε το καθήκον αυτό ταπεινά απλώς, να πάρετε όλη την εξουσία που σας δίνει, όλες τις δυνατότητε που σας δίνει η θέση αυτή. Και αν είναι να υποστηρίξετε κάποιους φακέλους, αυτός στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος ε, Ντιουρόν ε, για τους whistleblowers είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει και αν υπάρξει υποστήριξη από την κυβέρνησή σας, νομίζω ότι έχετε όλη τη δυνατότητα να Σημειώσετε σημαντική πρόοδο σε σημαντικά ζητήματα υπό τα δικαιώματα copyright όπως αναφέρθηκε και η συνάδελφος οι εκπρόσωποι της Προεδρίας στον τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό δεν ανέστηλαν την συνάντηση αλλά θα πρέπει να πιέσετε τα μέλη της Κορεπέρ να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, να καταλήξουμε σε ένα απτό αποτέλεσμα γιατί το Κοινοβούλιο επιθυμεί να έχουμε, να σημειώσουμε πρόοδο, να έχουμε ένα κείμενο συμπεφωνημένο. Νομίζω ότι η ιστορία, η μεγάλη ιστορία της χώρας σας και οι καλλιτέχνες τους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα σας δίνουν την ηθική δύναμη να πιέσετε να αναλάβετε όπως έλεγα όλοι σας την ε, αρμοδιότητα υπό την Προεδρία του Συμβουλίου για να προωθήσετε τους φακέλους αυτούς. Και να καταπολεμήσετε ίσως και τις πιέσεις που ασκούνται στο εσωτερικό της χώρας σας, ώστε να ξεπεράσουμε τα μπλοκαρίσματα που αντιμετωπίζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και εσάς κύριε Υπουργέ που είστε εδώ ε, για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Έχω αρκετά ερωτήματα γιατί εκπροσωπώ και άλλους τρεις συναδέλφους θα προσπαθήσω όμως να είναι όμως το δυνατόν πιο σύντομος. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η συνάδελφός μου η Λίδια Γκέριγκερ και ο συνάδελφος Ζαν ε, Μαρή Καβαντά. Η Ρουμανική Προεδρία, σε ό,τι αφορά το copyright, το δικαίωμα του δημιουργού, έχει την πρόθεση να κλείσει το θέμα μέσα στο εξάμεινο της, είναι ή όχι. Και συγκεκριμένα θα προσπαθήσετε να λύσετε στο δυνατόν λιγότερα, ε, πιο γρήγορα αυτό το ε, διέξοδο, ε, γιατί είναι επίγον να βρεθεί λύση. Και ασκούμε πίεση για σας, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και πραγματικά είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την όθηση που υπάρχει και να τελειώνουμε με το copyright. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ συλλογικές προσφύγε, τα συλλογικά ενδικά μέσα και τη σχετική οδηγία, πόσο μπορεί να προχωρήσει η Ρουμανική Προεδρία. Δεν θα υπάρχει άλλο τριμερής διάλογος σε αυτό το ε, εναπομένων ε, διάστημα. Ε, ουσιαστικά το Φεβρουάριο θα είχαμε τη δυνατότητα γιατί μετά δεν έχει άλλο ε, άλλη δυνατότητα, άλλο περιθώριο. Ε, θα μπορούσε να γίνει κάτι λοιπόν. Και το τρίτο στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά μου το έχει γράψει ο συνάδελφο, ε, ο Σάφο Ζάιρ συγκεκριμένα. Ο φάκελο ευθυγράμμισης επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αυτό το θέμα κρεμεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και ανεπίσημα η Κομισιόν μιλά για διάσπαση της πρότασης Omnibus. Οι γνωμοδοτούσε επιτροπέ και η δική μα επιτροπή θα ήταν υπέρ αυτή τη διάσπαση, του διαχωρισμού, για να έχουμε έτσι αυτά αποτελέσματα σε την ευθυγράμμιση πάνω από 60 νομοθετικών πράξεων ήδη. Και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι θα πρέπει να συζητηθούν και τα αναπομένοντα μέρη της πρότασης. Οπότε, αν μπορείτε, πείτε μα, εσεί αυτή την επιλογή πώ τη βλέπετε. Και αν μπορείτε να μα επιβεβαιώσετε την δέσμευση τη Προεδρία σα στο θέμα αυτό και παίρνω πάλι στα γερμανικά δύο ερωτήσει ε, προς τον Αφον Ντάνιελ Μπούντα και έχει να κάνει πιο πολύ τα εσωτερικά τη Ρουμανίας. Στα αγγλικά πάλι. Είστε μέλο κύριε Τάντερ, τη Επιτροπή Βενετίας. Ε, Πολλέ όμω από τι αποφάσει ε, αυτά τα διατάγματα τα επίγοντα δεν, που εκδώστε δεν είχαν ε, την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της ε, Βενετίας σε ό,τι αφορά το 1992 συγκεκριμένα, περσινά διατάγματα ε, και τα δύο αφορούσαν ε, την αλλαγή κάποιων νόμων για δικαιοσύνη. Δεν έχετε διαβουλευτεί την Επιτροπή ενώ δεσμευτήκατε να το κάνετε. Θα το κάνετε και γιατί δεν την έχετε ενημερώσει, ε, γιατί δεν έχει πληθεί και άλλων ε, τροποποίησεων δικαστικών ε, νομοθετημάτων. Και επίσης, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα με, δικαστικό μεταρρυθμίσεων με την έγκριση της Επιτροπής Βενετίας γιατί ε, δεν έχετε συμβουλευτεί την Επιτροπή της Βενετίας και αν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα το πράξετε από εδώ και πέρα. Πρωτού προβείτε σε άλλες μεταρρυθμίσεις, ε, αν έχετε χρόνο να θέσω και ένα άλλο ερώτημα το συνάδελφο Ντάνιλ Μπούντα. Πρόσφατα είπατε ότι έχει ένα επίσης κατεπήγον διάταγμα το Υπουργείο σας ε, σε σχέση με μια απόφαση του Ανώτατου Κυρωτικού Δικαστήριου ε, για την προσφυγή κάποιων ε, αποφάσεων ε, ώστε να κυρωθούν και να επαναδικαστούν υποθέσεις. Τι θα γίνει αν τα δικήματα που ενδεχομένως έχουν παραγραφεί θα ξαναγίνει δίκη ή δεν θα ξαναγίνει. Όταν μιλάμε για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, παραγράφεται το αδίκημα και τι γίνεται μετά. Πανέρχει, πρέπει να αποζημιωθούν ε, καθού. Και όταν υπήρξε κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πώς θα εξασφαλίσετε την προστασία των χρηματοπιστωτικών σφαίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, λέει στα γερμανικά πάλι. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Για μένα είναι πολύ σημαντικά τα δύο πρώτα ερωτήματα. Δηλαδή, δικαιώματα πνευματική ε, διοκτησίας, ε, και με τον Υπουργό δηλαδή, και το δεύτερο, συλλογικές, ε, συλλογικά ενδικά μέσα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Αυτά λοιπόν ήταν τα ερωτήματα που υπάβλαν τα μέλη. Α, δύο ακόμα λοιπόν ερωτήματα έχουμε. Η κυρία Χάουταλα. Ε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Ε, Υπουργέ, δεν είχαμε σαφή απάντηση από τους εκπροσώπους της Ρουμανικής ε, Προεδρίας σχετικά με τις συλλογικέ αποζημιώσεις που είναι ε, η βασικότερη πρόοδος για τα δικαιώματα των καταναλωτών υπό την ε, εντολή την παρούσα και θα ήταν απογοητευτικό να μην προχωρήσουμε. Ποια είναι τα σχέδιά σας σε αυτό. Δεν θα μπορούσατε να προχωρήσετε το θέμα αυτό, το φάκελο αυτό, στον κατάλογο προτεραιοτήτων σας. Δεύτερον, στα πλαίσια της δικαστικής σας μεταρρύθμισης και να σας πω ότι εμείς υποβάλλουμε τα ερωτήματα αυτά σε όλους τους εκπροσώπους των Προεδριών σχετικά με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση διαφθοράς είναι σημαντικό θέμα για εμάς γιατί θεωρούμε ότι το Συμβούλιο της Προεδρίας και γι' αυτό σας ρωτώ πρέπει να δίδει το καλό παράδειγμα. Ο κύριος Ποπά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η νομοθεσία σχετικά με τις ε, προσφυγές στο ανώτο δικαστήριο στο ακυρωτικό είναι κάτι αρκετά αμφίσιμο. Έχει συζητηθεί πολύ διότι το συνταγματικό δικαστήριο ήδη βρήκε περιπτώσεις παράνομης απόφασης του ακυρωτικού για την απόφαση 304 του 2004 σχετικά με το σχηματισμό των πενταμελών δικαστηρίων. Εάν αυτό είναι αληθές, σημαίνει ότι η Ρουμανία εκτός και αν αναλάβει μέτρα προς την κατέμψη αυτήν, θα διατρέχει τον κίνδυνο να παραπεμφθεί ε, στο δικαστήριο. από εκείνους που θα έχουν προσφύγει επί τη βάση των παρανόμως ε, σχηματιστέντων αυτών πενταμελών ε, δικαστηρίων. Πρόεδρος, έγιναν τώρα οι ερωτήσεις, αλλά εδώ κανονικά θα έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει ως προς το πρόγραμμα με το θέμα αυτό. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κύριο Υπουργό να απαντήσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Μία ώρα λέει ο Υπουργός. Όχι μία ώρα φοβούμε λέει ο Πρόεδρος κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές ε, μάλλον ε, δεν εμπίπτουν και στην αρμοδιότητά σας ως Υπουργού. Μπορείτε επ' αυτό να είστε και πάρα πολύ σύντομος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα καταφέρω να σας πείσω απολύτως. Αλλά εισαγωγικά ε, να πω ότι τα ερωτήματα που μου κάνατε διαρούνται σε δύο μεγάλες ομάδες. Ερωτήματα που απευθύνονται σε μένα ως προεδρεύοντος του Συμβουλίου Τζάι, ε, δικαστικών και εσωτερικών υποθέσεων και που μου απευθύνονται ως Υπουργό Δικαιοσύνη ω προ τι εσωτερικέ εθνικέ μα εξελίξει και όχι τη ευρωπαϊκή. Επαναλαμβάνοντας ότι βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Μάλλον θα έπρεπε να αποφύγω τη θεματική των εσωτερικών μας ζητημάτων στη Ρουμανία. Δεν θα το κάνω όμως αυτό. Δεν θα σας παραπέμψω στις εθνικές αρχές. Ως προς το κράτος δικαίου είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα. Μερικοί λένε ότι πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει κράτος δικαίου. Έχουμε κάποια στοιχεία, έχουμε κάποιες παραμέτρους που μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο περιεχόμενο της έννοιας αυτής, στον ορισμό αυτών. Και αναφέρομαι εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κράτος δικαίου πρέπει να συμμορφούνται προς τις συνθήκες, αλλά δομείται διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη, λαμβανομένων υπόψη των παραδόσεων, του παρελθόντος και φυσικά τις ιδιαιτερότητες των χωρών, των ανατολικών χωρών που βρίσκονταν υπό το κομμουνιστικό σύστημα. Κράτος δικαίου σημαίνει συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σημαίνει νομοθέτηση τηρώντας τις αρχές των ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων μη αναστρέψιμη και υπό τις κατευθύνσεις της ε, Επιτροπής της Βενετίας. Θα πω ότι δεν είναι συμπτωματικό ότι οι αποφάσεις των συνταγματικών δικαστηρίων είναι τελεσίδικες από την ημέρα της δημοσίευσής τους στην επίσημη εφημερίδα. και προσπαθώντας να απαντήσω το ερώτημα που εντέθη. Ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το κράτος δικαίου, γιατί δεν κάνει ισότιμες συστάσεις η Επιτροπή της Βενετίας προς τα κράτη-μέλη. Η απάντηση είναι ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές δομές. αλλά όλοι καλούμαστε να συμμορφωθούμε προς τις ίδιες ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα. Με ρωτάτε γιατί σε σχέση με τη διαταγή 92 την περισσυνή δεν προσαρμοστήκαμε προς τις... Ε, μάλλον γιατί δεν διαβουλευτήκαμε με την Επιτροπή της Βενετίας. Έγινε η διαβούλευση αυτό, αυτή. Ε, εγώ ο ίδιος πήγα στο Στρασβούργο τρεις φορές στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπή της Βενετίας, υπήρξα μέλος τα τελευταία πέντε χρόνια και η διαταγή 92 είχε έναν και μόνο σκοπό. Να αναλάβει υπό τη συστάσεις της Επιτροπής Βενετίας τα θέματα που δεν θα μπορούσαν και δεν θα έπρεπε να εξεταστούν διακριτά. Την απόσυρση των δικαστών μετά από 20 χρόνια ενεργού συμμετοχής. Δύο εκ των 5.000 δικαστικοί στην Ρουμανία ήταν έτοιμοι να συνταξιοτηθούν. Εκπρόσωποι λοιπόν της Επιτροπής Βενετίας και άλλων φορέων στην Ευρώπη εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι 2.000 περίπου δικαστικοί θα αποσύροντο το οποίο θα σήμαινε το 1 τρίτο του συνόλου των δικαστικών λειτουργών που είχαμε στη Ρουμανία. Επ' αυτού εγώ θα μπορούσα να υποβάλλω το εξής σχόλιο. Το να συνταξιοδοτείται ένας δικαστικός στα 45 χρόνια ηλικίας είναι κάπως πρόημο. Η σωστή λειτουργία του κράτους δικαίου ε, σημαίνει ότι ένας δικαστικός λειτουργός, ένας δικαστής στα 45 χρόνια ηλικίας, οπωσδήποτε είναι απολύτως σε θέση να συνεχίσει τη δουλειά του, τα καθήκοντά του, Πήγα εγώ τρεις φορές λοιπόν στο Στρασβούργο να συζητήσω το διάταγμα αυτό 92. Συζητήσαμε όλες τις δυνατότητες και πιθανές λύσεις. Συζητήσαμε και τις ε, περιπτώσεις πειθαρχικών κυρώσεων κατά δικαστικών λειτουργών, υπό τις οποίες θα έχαναν την δικαστική τους ανεξαρτησία υπό την, ε, στην περίπτωση μάλλον της υποβολής οποιασδήποτε κυρώσεως και υπό το διάταγμα 92 προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση ώστε τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών να, να μπορούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου. Εις τα δύο μέλη λοιπόν των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών εδόθη η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και αυτό απορρέει και από το Σύνταγμα. Έξι από τις συστάσεις της Επιτροπής Βενετίας ενσωματώθηκαν στο διάταγμα αυτό 92. Έχουμε τώρα τρία νομοθετήματα για τους δικαστικούς τα οποία έχουν τροποποιηθεί από το 1994 από το 2004 και εγώ πάντοτε επανέλαβα ότι είμαι απολύτως υπεύθυνος για τα όσα κάνω ή τα όσα λησμονώ ενδεχομένως αλλά όχι για αυτά που κάνουν άλλοι. Εδώ δεν είχαμε κάποιο έκτακτο διάταγμα, κάποια έκτακτη διαταγή. Η δικαστική νομοθεσία έχει επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Δεν μπορείτε λοιπόν να μου κάνετε την ερώτηση γιατί δεν διαβουλεύτηκα με την Επιτροπή όταν η νομοθεσία αυτή επικυρώθηκε. Πάντως, είτε με τη μορφή διατάγματος, είτε με τη μορφή νόμου, όλα αυτά τα νομοθετήματα ε, ελέγχονται και επικυρώνονται σύμφωνα με τη χρηστή κοινοβουλευτική και συνταγματική διαδικασία στη Ρουμανία. Πάω τώρα στο θέμα των whistleblowers. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στο φάκελο αυτό και δεν πρόκειται να κάνουμε καμία εξαίρεση για φορολογικά ή χρηματοδοτικά θέματα, χρηματοοικονομικά θέματα. Εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν υπέρ της, του περιορισμού του πεδίου για τις συλλογικέ αποζημιώσεις. Αυτό δεν είναι ένα θέμα αρμοδιότητος του Υπουργού Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Είναι θέμα ε, του Συμβουλίου Αντιογωνιστικότητας και είναι φάκελος που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, όπου θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright. Και αυτό δεν είναι θέμα Συμβουλίου Τζάι, αλλά είναι θέμα των αρμοδίων φορέων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εγώ ως υπουργό δεν είμαι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνη ε, πρέπει να διεκδικεί αρμοδιότητα επί οποιοδήποτε θέματος. Πρέπει να γνωρίζουμε την αρμοδιότητά μας και να λειτουργούμε εντός του πνεύματος και του γράμματος του νόμου. Καλή την πίστη. Και πάω στην τελευταία ερώτηση που μου απευθυνθήκε. Αναφερθήκατε στα έκτακτα διατάγματα και εκφράσατε μια ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία του κράτου δικαίου. Πρέπει να μας ανησυχούν και τα, οι περιπτώσεις δυσάρεστων για τυχόν κρουσμάτων, αλλά και τα όσα δεν κάνουμε προκειμένου να τα προλάβουμε. Ήδη τοποθετήθηκα ε, σχετικά με πιθανό ορισμό του κράτους δικαίου. Ε, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ως διαδικασία εφόσον εντοπίζουμε κάποια κενά ή κάποιες ελλείψεις και δεν αναλαμβάνουμε μέτρα ώστε να τις πληρώσουμε. συνέβη τα τελευταία 4-5 χρόνια να έχουμε αντιφατικές τοποθετήσεις μεταξύ διαφορετικών δικαστικών επιτροπών σχετικά με το σχηματισμό πενταμελών δικαστηρίων. Όταν όμως έχουμε τον ποινικό κώδικα που μας λέει κάποια στοιχεία τα δικαστικά συμβούλια ή οι επιτροπέ μας λένε κάτι διαφορετικό και διαφορετικές αρμοδιότητες με διαφορετικές περιοχές επικάλυψη, τα πράγματα περιπλέκονται. Και αυτά δεν τα λέει ο Υπουργό Δικαιοσύνη δηλαδή εγώ, αλλά τα λέει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Πάντως από την ευρωπαϊκή νομολογία αυτό που προκύπτει ε, ε, είναι ότι δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε ε, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη οποιοδήποτε πολίτη. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εισακουστούν από το δικαστήριο Και το οποιοδήποτε διάταγμα ή νομοθεσία εξετάζουμε δεν είναι προς το όφελος του α ή του β πολίτη, αλλά τις καλύτερης λειτουργίες του κράτους δικαίου. Όταν έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις, αυτές δεν μπορούν να καταργηθούν επί τη βάση του ότι το πενταμελές ή άλλο δικαστήριο που καταδίκασε δεν είχε την απαραίτητη αρμοδιότητα, για τελειώς θα διαταρασσόταν η ένομη τάξη. Και υπάρχουμε μάλιστα σημειώστε ότι έχουμε περισσότερες αθωωτικές παρά καταδικαστικές αποφάσεις από τα σχετικά αυτά δικαστήρια. Αλλά όλες οι αποφάσεις που θα έχουν εκδοθεί θα έχουν εκδοθεί επί τη βάση ε, διοικητικά επικυρωμένων αποδεικτικών στοιχείων. Δεν θα μπορούσαμε πάντως επί τη βάση της οποιασδήποτε σταθερότητας να παραβιάσουμε με συνταγματικές επιταγές. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλώ για το θέμα αυτό για μία ώρα και παραπάνω. Όλα τα σχετικά επιχειρήματα θα σας τα στείλω γραπτός και δεσμεύομαι. Ε, ε, έχω υπηρετήσει ως υπουργό για δύο χρόνια τώρα. Δεν είμαι μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος διορίστηκα υπουργό ε, μετά από θητεία δεκαετή στο συνταγματικό δικαστήριο. Δεν μπορώ λοιπόν να αγνοήσω τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου. Εφόσον κριθούν ένοχα συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά θα παραμείνουν υποκράτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που απαντήσατε στα ερωτήματα των βουλευτών. Σας εύχομαι και προσωπικά αλλά και στη Ουρβανική Περιφερεια εν γέννη καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και κύριοι. Ε, ευχαρίστω να ξαναέρθω όποτε με καλέσετε, όποτε με χρειαστείτε. Επιτρέψτε μου όμως να έχω περισσότερο χρόνο να μιλήσω για να μπορέσω να παρουσιάσω όλα τα επιχειρήματά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με, να συνεχίσουμε μάλλον με το σημείο 27 της ημέρης τη διάταξης. Ξεκινάει τώρα μια διαδικασία που έχει να κάνει με ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία ε, είναι ουσιώδη για τη λειτουργία ενός προτύπου SCP e στα αγγλικά και βεβαίως για το ίντερνετ, το διαδίκτυο των πραγμάτων. Πρώτα θα έχουμε μια παρουσίαση ε, μιας μελέτης που ζητήθηκε από το, το Γραφείο Πολιτικής ε, του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο πυρογνωμόνες και θα γίνει μια ακρόαση. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο το οποίο, για, τη, για την πνευματικά δικαιώματα που περιλαμβάνει μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό του SEP. Και τότε η Επίτροπος Μπιανκόφσκα μίλησε εδώ εν συντομία τον Ιούλιο του 2018. Σήμερα θα ακούσουμε πυρογνώμανες, οι οποίοι εξειδικεύονται σε ζητήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και θα μας πούν τι διακυβεύεται, ε, θα μας πούν ε, ε, το εξετάσουμε το θέμα από διάφορα, από διάφορα, από διάφορα οπτικές γωνιές. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την παρουσίαση της μελέτης αυτής. Ένας από τους συντάκτες, ο οποίος Λουκ Μακδόνα, ο οποίος ε, είναι καθηγητής ε, στο λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, είναι εδώ μαζί μας. Θα του δώσουμε το λόγο για 15 λεπτά περίπου. Έχετε το λόγο. Uh, it's a great honor to be here. I'm skip quickly on... Λοιπόν, θα, θα αφήσω την πρώτη ε, διαφάνεια. Πρόκειται για αυτή την έκθεση που αφορά το SCP και το διαδίκτυο των πραγμάτων που έκανα από κοινού με τον Ερνίκο Μπονάντιο. Ε, εξετάζουμε την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αναλύουμε, την, την ανακοίνωση τη 24 Νοεμβρίου του 2017 για το θέμα της τυποποίησης τεχνολογία και τα δικαιώματα των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Σα πω πρώτα δύο λόγια για το δεύτερο πλαίσιο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικά για να υπάρχει διαλειτουργικότητα. όπω το, το, το, τα 3G, 4G. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από οικονομική πλευρά, έτσι ώστε ε, να έχουμε οικονομίε κλίμακα, ε, να μπορούν τα προϊόντα να αντικαταστούν το ένα το άλλο, Τώρα με το διαδίκτυο των πραγμάτων και το big data, αυτό έχει να κάνει πλέον και με τα καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρικές συσκευές, ε, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, επίσης είναι ένας ε, τύπος ιδιοκτησίας που καλύπτει και μια σειρά από εφευρέσεις. Και αυτά τα, αυτές τις τεχνίες τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ένα πρότυπο ονομάζεται SCP. E και συχνά εκεί υπάρχουν και σημαντικές διενέξεις και διαφορές. Αυτές οι διαφορές μπορεί ορισμένες φορές να δημιουργήσουν εξαιρετικά προβλήματα, ε, σημαντικά προβλήματα συγγνώμη, στην παρασκευή, στην εμπορία και στην διανομή περίπλοκων προϊόντων. Ενισχύοντας τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι ιδιοκτήτες αυτών των SCP e μπορούν να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους ή να τους απαρεμποδίσουν ε, από την παραγωγή και την διανομή ε, αυτών των προϊόντων. Να μην τους αφήσουν, δηλαδή να το διαθέσουν στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ένταση μεταξύ των SCP e και των προτύπων. Θέλουμε να είναι η αγορά πιο δίκαιη, να υπάρχει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, να είναι πιο απλή πρόσβαση. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν στο κατάλληλο σημείο ισορροπίας. Μία απάντηση βεβαίως είναι να έχουμε δίκαιες πρακτικές σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Υπάρχουν οργανώσεις όπως η ΕΣΤΗ στην Ευρώπη που ζητούν οι ιδιοκτήτες να λαμβάνουν μια άδεια η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί και θα πρέπει βεβαίως να ακολουθούν τους κανόνες φραντ, δίκαιη, λογική, χωρίς διακρίσεις. Τι γίνεται όμως αν ο ιδιοκτήτης ε, και αυτοί οι οποίοι ε, θα έχουμε μελλοντικά τι άδειε, δεν συμφωνούν για το τι, τι εννοούμε με αυτά τα επίθετα. Τι μπορεί να είναι δίκαιο ή λογικό. Μπορεί κάποιο να θεωρεί ότι υπάρχουν διακρίσει ε, στους όρους ή μπορεί να υπάρχει διαφωνία σε ό,τι αφορά το εδαφικό πεδίο που θα καλύπτει η άδεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν διαφορέ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και για το ίντερνετ των πραγμάτων, διότι στο παρελθόν ο κατασκευαστή ενός smartphone, ενός laptop ήταν αυτός ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει τέτοιου ζητήματα. Τώρα όμως ε, υπάρχουν διάφορες ε, ηλεκτρονικές συσκευές ε, όπου μοιράζονται προσωπικά δεδομένα, τεχνολογίες με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Το να βρεθεί λοιπόν το κατάλληλο σημείο ισορροπία είναι κρίσιμη σημασία, είναι κρίσιμο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλέ διαφορέ για τα τα τη δικαστήριο η πιο διάσημη υπόθεση είναι η υπόθεση της Huawei. Ε, μετά από μια, ένα προδικαστικό ερώτημα φτάσαμε στο συμπέρασμα του δικαστήριο ότι δεν αποτελεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης για τον ε, ε, ιδιοκτήτη ενός ΣΕΠ να ε, κάνει μία, να ζητήσει μάλλον να, να κινηθεί κατά ενός ανταγωνιστή του εφόσον βεβαίως πληρεί συγκεκριμένε προποθέσει. Ποιε είναι οι υποχρεώσει, λοιπόν που πρέπει να πληρεί αυτός ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος αυτής της, της πρώτης για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει ε, κατάχρηση τη θέσης σύμφωνα και με τη συνθήκη. Ο κάτοχος ενός SCP, e ο οποίος έχει μια υποχρέωση FRAND, δηλαδή να δώσει μια άδεια με όρους FRAND, δεν μπορεί να ε, δεν οδηγείται σε δεσπόζουσα θέση ή σε, σε κατάχρηση αυτής εφόσον έχει ενημερώσει για την παράβαση των ενδιαφερόμενων και εφόσον κάποιος έχει δείξει ότι ετοιμάζεται να συνάψει μια συμφωνία και του έχει προσφερθεί γραπτός μια τέτοια συμφωνία, αναφέρονται εκεί όλοι οι όροι και η δεύτερη υποχρέωση που έχει ο, κάτοχος του SCP e είναι ότι το δίπλωμα βραστεχνίας ή μάλλον θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δίπλωμα αυτό που παραβαίνει την νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται δηλαδή στην προσφορά φραντ με βάση τις θεμητέ ε, εμπορικέ πρακτικές και την καλή πίστη. Ο κάτοχος λοιπόν του διπλώματο θα πρέπει να κάνει μια πραγματική προσφορά στον ανταγωνιστή του και εκείνο πρέπει να απαντήσει πραγματικά ε, σε αυτόν. Σύμφωνα βεβαίως με τι θεμητέ εμπορικέ πρακτικές, τις εμπορικές συγγνώμη. Εάν λοιπόν, ο ανταγωνιστή λοιπόν αυτό ο οποίο ε, παραβαίνει τον νόμο θεωρητικά, δεν ανταποκριθεί θετικά σε αυτή την πρόταση στα πλαίσια τη ΦΡΑΝ, τότε μπορεί να προσφύγει ο κάτοχο. Και εκεί δεν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσα θέση. Ε, δεν έχουμε ε, άλλε κατευθυντήριε γραμμέ, αν θέλετε, από αυτή την απόφαση. Δεν ξέρουμε πώ υπολογίζεται, παραδείγματο χάρη, το ποσοστό. Γι' αυτό τα εθνικά δικαστήρια που ασχολούνται με ζητήματα διπλώματα βραστεχνία καθημερινά έχουν πολλά ζητήματα που παραμένουν δυσεπίλητα. Έχουμε μια υπόθεση στον Ηνωμένο Βασίλειο αρκετά σημαντική ε, μετά την υπόθεση Huawei όπου το αγγλικό δικαστήριο ήταν διατεθειμένο να δώσει κάποιες σαφείς κατευθείας γραμμές για το τι αποτελεί φραντ στην περίπτωση αυτή. Στην αρχή είπε ότι μια παγκόσμια άδεια είναι φραντ, παραδείγματος χάρη. Ε, και το, είχε αποφασίσει να υπάρχει ένα ποσοστό, ένα benchmark για ένα τέτοιο ε, φραντ. Δίνονται λοιπόν ε, συγκεκριμένε κριτικέ γραμμέ στο δικαστήριο, οι οποίε ε, συμπεριλήφθησαν στην ανακοίνωση τη Κομισιόν, όπου λέγεται βεβαίω ότι πρόκειται για περίπλοκε υποθέσει που πρέπει να επιλύονται αναπερίπτωση. Στην έκθεση επίσης εξετάζουμε γερμανικές, γαλλικές και αγγλικές υποθέσεις, στα δικαστήρια αυτών των χωρών δηλαδή, πριν από μερικού μήνε είχα μια απόφαση στη Γερμανία για το θέμα του κατά πόσο κάποιο ο οποίο έχει αγοράσει ε, ένα SCP e ε, δεσμεύεται από τι πρώτερε ε, υποχρεώσει φραντ που είχε ο προηγούμενο ε, ιδιοκτήτη. Και από ό,τι φαίνεται εκεί το δικαστήριο λέει ότι ο δεύτερο αυτό ιδιοκτήτη δεσμεύεται. Τι λέει τώρα η ίδια η ανακοίνωση. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η έμφαση στην διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόλυτη ενημέρωση για τα πρότυπα αυτά και για τα διπλώματα βρετεχνία και αυτέ οι πληροφορίε ε, όχι μόνο είναι ατελεί, αλλά δεν είναι και εύκολα προσβάσιμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ένωση, μεταξύ των οργανώσεων που θεσπίζουν τα πρότυπα, όπω η ΕΣΤΗ και βεβαίω ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλώματα Βρετεχνία. Ε, υπάρχει μια μόνη γνωμόνων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό όλα αυτά τα θεσμικά όργανα, όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να εργαστούν πιο σκληρά. Ε, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πληροφοριών που υπάρχουν ε, και μεγαλύτερη συμφωνία όλων αυτών των φορέων για να είναι πιο προσβάσιμη αυτή η πληροφορία. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση αυτών των ΣΕΠ, η γενική αρχή που, λέει, που αναφέρει η έκθεση ε, στην ανακοίνωση μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υγιή. Καλή πίστη, αξία της αγοράς για την τεχνολογία, ε, το, το προσδοκόμενο ζωή αυτή τη άδεια κλπ. Ε, όμως, όπως φάνηκε και στην υπόθεση Huawei και στον έγγραφο τη Κομισιόν, υπάρχει έλλειψη λεπτομερών στοιχείων για το πώς θα καθοριστεί το κατάλληλο ποσό ανάλογα με την περίπτωση η ανακοίνωση δεν λέει πολλά πράγματα επ' αυτού. Αναφέρονται απλώς κάποιες γενικές αρχές. Κάποιοι επέκριναν την ανακοίνωση ε, της Κομισιόν, διότι δεν δίνουν περισσότερα στοιχεία. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις περιπτώσεις και στην έκθεση και εμείς συμφωνούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει εκεί να έχουν ένα περιθώριο ελιγμών, είναι περίπλοκες περιπτώσεις και η προσέγγιση αναπερίπτωση ίσως είναι ένας πιο δίκαιος τρόπος για να επιτευχθεί το σωστό σημείο ισορροπίας. Υπάρχουν ε, όμως κάποια ε, επιχειρήματα στην έκθεσή μας ε, που σίγουρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση. Οι κάτοχοι του SCP e πρέπει ε, να αναφέρουν στο μέτρο του δυνατού ποιοι είναι οι όροι της, α, της άδειας. Ε, φορές ε, ε, δεν δίνονται καθόλου τα στοιχεία αυτά για ένα SCP. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Οι οργανώσεις οι οποίες θεσπίζουν τα πρότυπα θα μπορούσαν παραδείγματο χάρη να έχουν ένα σύστημα ε, πληστηριασμού για να βρουν την καλύτερη δυνατή τεχνολογία πριν γίνουν πρότυπα συλλογική, συλλογικές άδειες επίσης ε, είναι μια λύση και βεβαίως οι πλατφόρμες ε, open source για να αυξηθεί η διαφάνεια. Επίσης στην έκθεση θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο ισορροπημένη εφαρμογή ε, έχει τη σημασία της πέρα από την προσέγγιση αναπερίπτωση και την επικέντρωση και την επικεντρωθούμε στην εθνική νομοθεσία ε, υπάρχουν και άλλες λύσεις υπάρχουν μέθοδοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου ζητήματα όπως τι τις υποθέσεις Φραντ το δικαστήριο ε, θα έχει ένα ε, διατητικό όργανο που θα ασχολείται μόνο με αυτά τα ζητήματα υπάρχουν λύσεις διαμεσολάβησης στα συμπεράσματα λοιπόν τα συμπεράσματα είναι κατάλληλα, είναι τα σωστά γενικά αυτά της, της για τη διαφάνεια ε, και για τη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται για να έχουμε καλύτερη πληροφορία, καλύτερη πληροφόρηση αυτών που εφαρμόζουν τι τεχνολογίε αυτέ που καλύπτονται από αυτά τα SCP. E Θα πρέπει να βαστούμε σε κάποιε γενικέ αρχέ, την καλή πίστη, ε, το, τις λογικές ε, προσδοκίες ό,τι αφορά την αξιολόγηση και βεβαίως ό,τι αφορά την εφαρμογή που συνδέεται με την αξιολόγηση η αναπερίπτωση προσέγγιση φαίνεται λογική να εξετάζονται και εξετάζω βεβαίω την την, ποικιλομορφή, την ε, διαφορετικότητα των συνομολογίας είναι επίσης λογικό αυτό. Θα πρέπει τα SCPs e ε, να κοινοποιούνται, υπάρχουν οι άλλες ιδέες τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, όπως τα οι πλατφόρμες open source, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Αυτό ολοκληρώνει την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να την παρουσιάσω εδώ σήμερα και τώρα δίνω ξανά το λόγο στον Πρόεδρο. Ε, thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε και ελπίζουμε θα παραμείνετε μαζί μας διότι ακολουθεί ακρόαση για το θέμα αυτό και ενδεχομένως υπάρξουν ερωτήσεις από τους βουλευτές. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, όλες αυτές τις απαντήσεις ε, να τις ακούσουμε στο δεύτερο τμήμα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 28 που είναι η ακρόαση για το ίδιο ακριβώς θέμα. Θέλω να καλωσορίσω δύο μιλητές καθηγητή Ρούντι Μπέκερς, που είναι πρόεδρος ε, για τα θέματα τυποποίησης ε, ε, νοητικής ιδιοκτησίας, πρόεδρος της ομάδος της για τεχνολογία, καινοτομία, κοινωνία και στο Πανεπιστήμιο του Χόβεν στο τμήμα μηχανικής, μηχανικής και καινοτόμων επιστημών και έχουμε μαζί μας τον Μιχαήλ Φρόλινγκ που είναι διευθυντής ε, σε θέματα ευρωπαϊκών διεθνών νομικών υποθέσεων από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Νομάτων Εύρεσης Τεχνίας. Ε, κύριε Μπέκερς, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας σήμερα επειδή έχετε εκτεταμένη εμπειρία για το θέμα θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας ακαδημαϊκή προσέγγιση και άποψη και έπειτα θα λέω τον κύριο Φρέλιχ. 15 λεπτά έχετε κύριε Μπέκερς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να έρθω εδώ και να συζητήσουμε μαζί. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συντάκτες της μελέτης. Πάρα πολύ καλή η μελέτη, διότι παρουσιάζει και με συνοπτικό έβλεπτο τρόπο το τι συμβαίνει στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Εγώ είχα ετοιμάσει την παρουσίασή μου προτού διαβάσω τη μελέτη του προαλήσαντος, οπότε ίσως υπάρξουν κάποιες αλληλεπικαλύψεις και επαναλήψεις. Θα ήθελα να σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για τα, ε, τη σχέση αυτή μεταξύ διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και προτύπων και τι προβλήματα ανακύπτουν. Να μιλήσω για το μηχανισμό που έχουμε, θα τον έλεγα ένα μηχανισμό αυτοδιαχείρισης. Θα μιλήσω για τους πιθανούς ρόλους των αρχών και των ρυθμιστών, ιδίως ε, από δημόσια σκοπιά. Θα σα εξηγήσω γιατί έχουμε τόσο μεγάλε εντάσει την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα θέμα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντιπαράθεση. Θα δούμε του διάφορου εμπλεκομένου φορεί, όχι μόνο τον ακαδημαϊκό κλάδο, αλλά και τη βιομηχανία, τι προκλήσει έχουμε στην Ευρώπη για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, ΜΜΕ και βέβαια ε, τι ε, προκλήσει για την κοινωνία και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τεχνικά πρότυπα. Μπορεί να μην γνωρίζουμε όλοι τι είναι, πάντως είναι τεχνικά, τεχνολογικά η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας. Βλέπετε στην οθόνη ε, αυτές τις διαφάνειες. Ε, αυτό χρειάζεται τη CPIP, format ε, γράφων. Δεκάδες πρότυπα χρησιμοποιούνται για να δείτε εσείς αυτή τη διαφάνεια που πολλές φορές μπορεί να μην είναι ορατά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τις κοινωνίες μας. Και σε λίγο θα σας εξηγήσω τι θα γίνει για τις επόμενες δύο-τρει δεκαετίες. Θα είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά τα πρότυπα. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή τη μεγάλη παράθεση. Αυτό ε, έρχεται και στο επόμενο, ότι και η τυποποίηση και τα διπλώματα ευρεσιτεχνή έχουν ως στόχο την καινοτομία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ε, και αυτό γίνεται με συμπερίληψη, με ένταξη από την πλευρά των ε, ε, προτύπων. Αλλά από την πλευρά των διπλωμάτων έχουμε την αντίθετη διαδικασία, εξαίρεση. Ε, δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει κάποια εφεύρεση. Προσπαθούν δηλαδή τον ίδιο στόχο να επιτύχουν, αλλά η σχέση μεταξύ τους δημιουργεί πρόβλημα πολλές φορές. Είπα και ο προλαλής σας, ότι έχουμε αυτά τα SCPs, αυτά τα ουσιώδη για τη λειτουργία συγκεκριμένου προτύπου ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και επομένω οι κάτοχοι ενό ΕΠΕ έχουν μεγάλη εξουσία στα χέρια του. Και δεν μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση στην αγορά αν δεν έχει ε, πρόσβαση αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Ε, δεν μπορεί να κάνει κάποιο μια άλλη επιλογή. Ο ανταγωνιστή δεν έχει περιθώρια και βέβαια πάρα πολύ λογικό να πάρει κάποιος ένα τέτοιο ΣΕΠ ε, και ως διαπραγματευτικό ατού μπορεί να υπάρξει η διάθεση στο εμπόριο κτλ. Και γι' αυτό βλέπουμε αυξάνεται ο αριθμός αυτών των προτύπων. Μπορεί να ήταν το δεκαετία 90 ε, κάποιες δεκάδες χιλιάδες, τώρα πάνω από 250 χιλιάδες. Αυτά τα ε, διπλώματα που θα μπορούσαν να είναι ουσιώδη για κάποιο πρότυπο, να είναι ΣΕΠ δηλαδή. Τώρα τα χρειαζόμαστε ναι ή όχι. Ε, πρέπει να πω ότι υπήρχαν ε, πρότυπα πάρα πολύ καλά που δεν κατοχυρώθηκαν με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Μπορεί να ήταν ε, ελεύθερη η τεχνολογία. Δηλαδή δεν υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνία πάντοτε, τα οποία είναι και εμπορεύσιμα για όλα αυτά τα πρότυπα. Γιατί θα θέλαμε κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνία συνδέεται με κάποιο πρότυπο. Γιατί θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό πρότυπο και θέλω να δώσουμε κίνητρα στο να μπορούν να συμμετέχουν στη βελτιστική τεχνολογία, αν μπορούν να περιλάβουν αυτήν την ε, τεχνολογία προτύπων. Το θέμα βέβαια είναι το κόστος να είναι μικρότερο του κέρδους. Τι είδους ε, φόβοι υπάρχουν όταν μιλάμε για το, τη σχέση αυτών των δύο πραγμάτων και την πολυπλοκότητα ή την αντιπαράθεση μεταξύ του. Πρώτον, είπαμε ότι όποιο έχει αυτή τη τεχνολογία έχει και εξουσία στα χέρια του. Τι μπορούμε να ε, φοβόμαστε. Λοιπόν, τη μη θεσιμότητα. Δέκα χρόνια εργαζόμαστε για να δούμε τελικά ότι δεν υπάρχουν ε, για διοδότηση βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ξαναξινάμε από το μηδέν. Αυτός ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνία μπορεί να ζητήσει πολύ μεγαλύτερη αποζημίωση αμοιβή, αφού συμπεριληφθεί σε ένα πρότυπο από όταν μπορούσε να έχει διαπραγματευτεί πριν. Δηλαδή αυξάνεται ε, η πίεση που μπορεί να έχει και γίνονται και ακαδημικές συζητήσεις και στη βιομηχανία για το πόσο μεγάλο μέγεθος μπορεί να έχει, να έχει αυτή η νέα εξουσία. Ακόμη και βραβεία Νόμπελ έχουν γράφει, έγγραφα που δείχνουν ότι πιστεύουν σε αυτό το μηχανισμό και ε, ότι υπάρχουν πιθανά προβλήματα. Μπορεί να ε, ε, συγκεντρώσουν επίσης όλα αυτά τα τέλη και επίσης μπορεί να μην υπάρχει και δίκαιη κατανομή και υπάρχει και το κόστος ε, συναλλαγής, όλα αυτά θα πρέπει να τα διαπραγματευτούν. Υπάρχει αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά επιχειρηματικά σχέδια, αν αναπτύξει μια ΜΜΕ, ε, μια τεχνολογία, αλλά δεν ξέρει ποιο θα χτυπήσει την πόρτα, ποια θα είναι τα θεμητά αιτήματα, πώ αυτά θα συνυπολογιστούν στην τιμή του προϊόντος κτλ. Έτσι, μπορεί να αυξηθούν οι τιμέ, να μειωθεί ο ανταγωνισμό. Ε, η παροχή ε, προϊόντων, άρα λιγότερα τα κίνητρα τελικά για τον καταναλωτή και τον Ευρωπαίο πολίτη, ανάλογα με το τι θα γίνει στο τέλος. Άρα δεν είναι καινούργια αυτά που σα λέω τώρα. Για πολύ καιρό έχουν απασχολήσει όλου. Και όταν τα έγραφα όλα αυτά, έφτασα και μέχρι τη δεκαετία του 1930, όταν πρώτο ξεκίνησαν οι οργανισμοί τυποποίηση και αναγνώρισαν και την αρχή και το πιθανό πρόβλημα αυτή τη μονοπολιστική τάση, όπω την ονόμασαν, και σκέφτονται τι μπορούμε να κάνουμε ήδη από τότε. Και χρειάστηκαν πολύ περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, στη δεκαετία του 1990 πρώτο θεσπίστηκαν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Τι έγινε λοιπόν στη δεκαετία του 90, κινητή τηλεφωνία, το GSM ε, όπως το ξέρουμε, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη. Τεράστια επιτυχία. Όχι για όλους όμως. Διότι τελικά υπήρξαν προβλήματα με διπλώματα ευρεσιτεχνία και πολλές μικρομεσαίε επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην αγορά αυτή. <coughs> Πολλές δε μεγάλες επιχειρήσεις είχαν εξ, επίσης αποκλειστεί. Δεν υπήρχαν ε, κάποιοι κανόνες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και έτσι καθαρίστηκε ότι χρειάζονται κανόνες και αρχές και μπήκαν ιδίω σε βασικούς αρχούς ανάπτυξης προτύπων αυτοί οι κανόνες. Γι' αυτό μιλάω για αυτοδιαχείριση. Αποφάσισα κάποιοι να ε, υιοθετήσουν πολιτικές όπως αυτές τι πολιτικέ φράντα που είπε ο που έχουν σχεδόν όλες τώρα οι οργανώσει ανάπτυξη προτύπων ε, διαφέρουν σε διάφορε πτυχέ, και, ε, υπάρχει μια ποικιλομορφία, αλλά υπάρχει και συζήτηση για το κατά πόσο να είναι επαρκεί κανόνε αυτοί, αν χρήζουν διευκρίνηση, επιμέρωση, επικαιροποίηση. Όλα αυτά τα συζητούν και οι ίδιοι φορεί. Τι είναι το φράντα και αυτοί οι κανόνες. Ως εξής λειτουργεί το πράγμα. Υποχρέωση για όλους, όλα τα μέλη να ενημερώνουν ε, αν θεωρούν ότι έχουν πιθανώς ουσιώδη διπλώματα ευρεσιτεχνής για τη λειτουργία ενός προτύπου. Έπειτα θέλουμε να ε, ζητηθεί ε, από αυτούς τους κατόχους να δεσμευτούν ότι θα διοδοτήσουν αυτά τα ΣΕΠ με τρόπο φραντ, δηλαδή δίκαιο, λογικό και μη διακριτικό και πρέπει να το σέβονται αυτό. Δηλαδή η τεχνολογία τους πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε έξι δις ε, συσκευές, ε, μηχανήματα. Για ε, άρα τη δέχονται τη συμφωνία οι εταιρείε από το να, αντί να κινδυνεύσουν να μην διατεθεί πουθενά η τεχνολογία τους σε καμία συσκευή. Έπειτα υπάρχει η διαπραγμάτευση της άδεια, διμερός ίσως ή συλλογικά μέσω των λεγόμενων δεξαμενών διπλωματών ευρεσιτεχνία. Και αν υπάρξει κάποια διαφορά, τελικά υπάρχουν εξοδετεμένα δικαστήρια που θα κρίνουν αυτή τη ε, δικαστική διαφορά. Δεν παίζουν ρόλο οι οργανισμοί ανάπτυξη προτύπου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εφαρμογή τη τεχνολογία, κάποιοι λένε ότι με τέτοιου είδου μηχανισμούς ε, έχουμε και το αντίθετο από το λεγόμενο hold out, ότι μια εταιρεία δεν παίρνει καν την άδεια, επειδή γνωρίζει ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνε. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τη δούμε αλλιώ ε, την όλη υπόθεση, με κάποιες αποχρώσεις. Πολλοί θεωρούν πάντως ότι υπάρχει και το αντίθετο ε, αποτέλεσμα, hold out δηλαδή που δεν πληρώνεται, δεν θέλω να πληρώσω. Τώρα, τι γίνεται από την πλευρά των διαφόρων αρχών και ρυθμιστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει διάφορα. Έχει ξεκινήσει κάποιε μελέτε. Δημιούργησε ευαισθητοποίηση, υπήρξε διάλογο για το θέμα. Θα τα πω και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Υπήρξαν και διάφορε δημόσιες διαβουλεύσει με πάνω από 100 stakeholders ε, και 2.000 σελίδε σχόλια. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η αρμόδια για την ε, πολιτική ανταγωνισμού δραστηριοποιείται και σε διάφορες τέτοιες υποθέσεις, συμμετέχει ε, στη, συμβουλευτικά στο πλαίσιο των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων, συμμετέχει στις συζητήσεις, όπως είπα, υπάρχουν και κάποια έγγραφα πολιτικής, ανακοίνωση κομισιών που μας είπε ε, ο προλαλής σας. Επίση, συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση, εκφράζει απόψει κομισιών και πολλέ φορέ μιλά και για κάποιου ασφαλεί λιμένε για τη συλλογική αδειοδότηση. Όπω οριζόντιε κατευθυντήριες γραμμέ, οι λεγόμενε πράσινε επιστολέ green letters. Και βέβαια έχουμε και το δικαστικό σύστημα, τα εθνικά δικαστήρια και βέβαια αυτά έχουν την τελευταία λέξη σε τέτοιου είδου διαμάχες. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο πολύ τι λένε οι διάφορε μελέτε που έχουν διεξαχθεί. Δεν θα επεκταθώ σε όλε, αλλά προσφέρουν πολύτιμο υλικό που το έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αναθέσει αυτές τις μελέτες που μας ε, εισάγουν στο θέμα, εκτιμούν και μελετούν τα διάφορα ζητήματα, ανοιχτέ πηγές, διακυβέρνηση. Τις βλέπετε, εγώ συμμετείχα σε δύο-τρεις μελέτες ε, και θα ήθελα να τονίσω μία από αυτές που νομίζω ότι έχει σημασία και στη σημερινή συζήτηση, η λεγόμενη ε, μελέτη περί αναγκαιότητας ή essentiality. Γιατί είπα ότι υπάρχει αυξανόμενη ένταση. Φαντάζομαι δεν σας διέφυγε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, ε, δίκες ε, και συζήτηση στη δημόσια κοινή γνώμη για αυτά τα ΣΕΠΑ. Υπάρχει ένας λόγος πόλεμος μεταξύ προτύπων διπλωμάτων ευαισθητεχνίας. Σχεδόν σε όλα τα δικαστήρια υπάρχει μια τέτοια υπόθεση. Άρα πρέπει να ρωτήσουμε αυτές οι δίκες, οι δικαστικές υποθέσεις μας ικανοποιούν, σημαίνει ότι λειτουργεί καλά το σύστημα και εργάζεται και το δικαστήριο σωστά ή βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου, άρα δεν είναι μεμονωμένες ε, και διάσπαρτες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει εν γέννη ένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι ομαλός ο, οργανισμός, ο μηχανισμός αδειοδότησης, λειτουργεί αυτή η βλεπουμε την κορυφη του παγοβουνου αρα δεν ειναι μεμονωμενες και διασπαρτες περιπτώσει, αλλα υπαρχει εν γεννη ενα προβλημα δηλαδη ειναι ο οργανισμος ο μηχανισμος αδειοδοτησης λειτουργει αυτη η αγορα και επειδή συμμετείχα σε πολλέ από αυτέ τι υποθέσει, γιατί ήμουν εμπειρογνώμων, πραγματογνώμων μάρτυρα, πρέπει να πω ότι ε, η αγορά αδειοδότηση έχει κάποια προβληματικά στοιχεία, μάλλον δεν είναι μόνο, ε, δεν είναι μονομένα όλα αυτά. Και είναι τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους εμπλεκομένους φορείς και τη βιομηχανία. Σε ορισμένα έχει αναφερθεί ανακοίνωση επιτροπής. Ε, επειδή δεν μπορούσα να φέρω ένα μακροσκελέστα το κατάλογο εδώ, έχω κάνει μια επιλογή. Μια, ένα από τα θέματα λοιπόν είναι αν αυτό το εύλογο τέλος θα πρέπει να σχετίζεται με τις τουρκικές δυνατότητες ε, ή με κάποιες από αυτές. θα πρέπει να δούμε την ε, λιγότερη, τη μικρότερη μονάδα, το τσίπ, τον υπολογιστή ή να δούμε το προϊόν συνολικά, αν είναι ένα αεροπλάνο, ξέρω εγώ, που είναι ακραίο παράδειγμα. Για να οριστούν λοιπόν τα τέλη και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς διαφοροποιούνται οι αγορές και εφαρμογέ από τον κάτοχο. <coughs> η ίδια αξία του προτύπου ή μάλλον του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται ή και ανάλογα της αγοράς ή όχι. Ένα άλλο. Ε, Ποιο εξουσιοδοτείται στην αλυσίδα αξία, ο τελικό χρήστη, η τελική συσκευή, ο τελικό χρήστη του αυτοκινήτου, του ε, τηλεφώνου κτλ. κτλ. Ή όχι. Ένα άλλο θέμα είναι η πληροφόρηση και διαφάνεια. Το είπε και προλαλή σα. Πολλά θέματα βέβαια. Πολλές, πολλά διπλώματα αυτή τη στιγμή. Θεωρούνται δυνητικά ουσιώδη, αλλά έχουμε 250.000 πρότυπα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι, μάλλον διπλώματα, ποια είναι ε, ουσιώδη για την και ποια δεν είναι. Και υπάρχει ασημέτρια πληροφόρησης αυτός που εφαρμόζει, αυτός ε, που εκτελεί, έχει λιγότερες πληροφορίες στη διάθεσή του. Και μιλάμε για το μηχανισμό της μη διακριτική μεταχή μεταξύ των προτύπων. Μπορεί κάποιος να ελέγξει. Άρα πολλά είναι τα στοιχεία. Κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς σίγουρα, αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες ε, σημαντικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και όπου να είναι θα ολοκληρώσω, αν μου δίνει ένα λεπτό ο πρόεδρος, για την Ευρώπη, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι σημαίνουν όλα αυτά και για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τι προκλήσει κοινωνία πρέπει να δούμε μαζί με αυτό το διαδίκτυο των πραγμάτων. Στην Ευρώπη συνολικά αντιμετωπίζουμε μεγάλε αλλαγέ ενέργεια, κινητικότητα, ασφάλεια, υγεία, ευημερία, τεχνολογίες φυσικά. Έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Είμαι και από τεχνολογικό πανεπιστήμιο και τα λέω και τα παραδέχομαι. Αλλά και ε, θετικά πράγματα μπορούν να φέρουν τεχνολογίες, ευφύες τεχνολογίες. Ε, Παραδείγματο χάρη ηλεκτρονική υγεία, τη βιομηχανία 4.0, το διαδικτυό πραγμάτων. Όλα αυτά τα λέω γιατί μιλάμε εδώ για πρότυπα και δεν είναι απομονωμένα, λειτουργούν μαζί όταν είναι συνδεδεμένα, υπάρχει, όταν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Άρα τα πρότυπα σε αυτές τις αγορές παίρνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό λοιπόν είναι και τόσο σημαντική σημερινή συζήτηση. Η μελλοντική αγορά που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη χρειάζεται πρότυπα και καλές υποδομέ και μηχανισμούς. So as a result, there will be a dramatic increase and change in... Θα έχουμε δραματικές αλλαγές ε, στον κλάδο Και δεν θα περιορίζεται στην κινητή τηλεφωνία. Στο μέλλον σε διάφορε εταιρείε, αλυσίδε αξίας, ε, αγορές, ε, από αυτοκινητοβιομηχανία, κοινωνική ε, υγεία κτλ. Τομεί που πριν δεν ε, λαμβάνονταν υπόψη. Θα επεκταθεί πολύ το πεδίο. Χρειάζεται γνώση, αλλάζει ο κλάδος και στην Ευρώπη για μένα είναι σαφέ ότι και οι ΜΜΕ έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν το πλαίσιο αυτών των αλλαγών που είπα. Αλλά θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Ε, και τέλο, θέλω να πω ε, ότι χρειάζονται ομαλοί ε, κανονισμοί αδειοδότηση λόγω των αλλαγών αυτών. Η Κομισιόν ε, έχει αναφέρει στην ανακοίνωσή τη, για παράδειγμα, τη διαφάνεια Υπάρχει κάποια, αλλά θέλουμε περισσότερη, κάποια καθοδήγηση για το τι είναι λογικό και δίκαιο. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Καλύτεροι μηχανισμοί, πιστεύω, από την έννοια τη μη δεκτική μεταχείριση, πολύ ωραία η αρχή, η μη διάκριση, αλλά δεν ξέρει κανεί αν δεν έχει πιο πολλά στοιχεία, αν υπάρχει δεκτική μεταχείριση προώθηση εναλλακτικών μηχανισμών όπω αυτέ οι δεξαμενέ διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για όλου όσου δραστηριοποιούνται στην αγορά και τα καταφέρουμε όλα αυτά τα επόμενα χρόνια θα είναι προ το όφελο όλων. Και αυτών που εφαρμόζουν και, από, και για αυτού που εφαρμόζουν του implementers και για αυτού που είναι καλόπιστοι κάτοχοι ενό ΣΕΠ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Professor, for this very important. Σας ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική αυτή εισήγηση, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φρόλιχ, επίσης για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι, εδώ μαζί σας ε, και έχω την ευκαιρία σήμερα να σας κάνω αυτή την παρουσίαση την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πολύ σύντομη εισαγωγή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρωστηχνίας. Είναι ένας από τους προγόνους της δομής των, ε, της προστασίας διπλωμάτων ευρωστηχνίας στην Ευρώπη. Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός επί τη βάση της ε, Σύμβασης Διπλωμάτων ευρωστηχνίας για την Ευρώπη Είμαστε, αν θέλετε, το εκτελεστικό σώμα του φορέα, του οργανισμού. Έχουμε 7.000 ε, υπαλλήλου, ε, εκ των οποίων 4.500 ανθρώπους που εξετάζουν τις υποβολές για διπλώματα, <clears throat> προκειμένου να καταλήξουν στο κατά πόσο θα πρέπει να παραχωρήσουμε δίπλωμα ή όχι στην συγκεκριμένη εφεύρεση. Η EPO διαδραματίζει όλο και με πιο σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση και στο ρόλο που διαδραματίζουν τα τεχνικά πρότυπα εδώ. Έχουμε πάρα πολλές επικαλύψεις αλλά και τριβή πολύ συχνά και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μία προσέγγιση μετά από 15 χρόνια συνεργασίας με διάφορους φορείς ε, ε τυποποίησης προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των διπλωμάτων και να αυξήσουμε και τη διαφάνεια. Ιδιαίτερα των ε, ουσιοδών διπλωμάτων των SCP. Μαζί με τον φορέα έτσι σχετικά ε, με τα SCP έχουμε αναπτύξει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που αφορούν και στην εργασία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και τη ΣΕΝ και ΕΛΕΚ που είναι οι άλλοι δύο φορεί τυποποίησης που είναι σημαντικοί εδώ, προκειμένου να προχωρήσουμε προς την ψηφιακή κοινή αγορά και ε, τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Επίσης έχουμε προεκτείνει την ε, λειτουργία μας για να συμπεριλάβουμε και άλλους σημαντικούς ε, οργανισμούς, το ITU-T, το IEC και το IEEE-SA μεταξύ άλλων. Η προσέγγιση μας είναι να ε, χρησιμοποιούμε έγγραφα σχετικά με τα πρότυπα. Θα πρέπει να έχουμε εντοπίσει πρακτικές και τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται όταν εξετάζουμε υποβολές διπλωμάτων ή Υπό την σύμβαση πνευματικής ιδιοκτησίας <clears throat> πρέπει μια εφεύρεση να είναι καινούρια και, δηλαδή, είναι καινούριο ένα δίπλωμα αν δεν θεωρείται εμπίπτη, ότι εμπίπτει στις τεχνικές ε, που σημαίνουν ότι διατίθεται μία συσκευή ή μία τεχνολογία στο ευρύ κοινό ήδη. Τώρα αυτά μαζί με τους οργανισμούς τυποποίησης είναι ένα πολύ σημαντικό πλέγμα πλαίσιο ε, εγγράφων και στοιχείων, όπως και προκατακτικών σχεδίων και άλλων ε, στοιχείων κοινοποίηση προηγούμενης ενημέρωσης που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στις υποβολές τους ή να λαμβάνονται στα πρακτικά των συναντήσεων αυτών. <coughs> Στη διαδικασία αυτή ανάπτυξης ε, προτύπων όλα αυτά μπορούν να είναι ε, κοινοποιήσιμα για το ευρύ κοινό εκτός αν έχουμε διατάξει εμπιστευτικότητος. Αυτά δεν είναι πάντοτε δυνατά για την ΕΠΟ γιατί οι περισσότεροι οργανισμοί τυποποίησης διαχέουν τα έγγραφα αυτά μόνο στα μέλη τους. Αναγνωρίζοντας την σημασία των εγγράφων αυτών, των αποδεικτικών αν θέλετε αυτών εγγράφων και αναγνωρίζοντας ε, την ανάγκη να έχουν την υψηλότητα τη δυνατή ποιότητα, έχουμε ε, συνάψει ε, συμφωνίες συνεργασίας με διάφορους ε, οργανισμούς πιστοποίησης ώστε να, τυποποίησης ώστε να λάβουμε τα αποδεικτικά τους έγγραφα ώστε να παραχωρούμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας μόνο για εφευρέσεις που είναι πραγματικά καινοτόμες και όχι τεχνολογίες που ήδη είναι κοινοποιημένε, είναι γνωστές δηλαδή στην κοινή γνώμη. Η συνεργασία αυτή μεταξύ της ΕΠΟ και των STOs, δηλαδή των οργανισμών τυποποίησης, είναι γνωστή στα μέρη και στους υποβάλλοντες και μας βοηθάει να βελτιστοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα και την διαφάνεια των διπλωμάτων. Επίσης μας βοηθάει να μειώσουμε επακθή ε, διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε την αύξηση Ε, της ποσότητας των εγγράφων ε, τυποποίησης που λαμβάνουμε από τους διάφορους STO που είναι άνω των 2 ε, εκατομμυρίων έγγραφα το 2017 και υποβάλλονται προς τους υπευθύνους εξέτασης της EPO οι οποίοι επίσης τακτικά διαβουλεύονται, συμβουλεύονται μάλλον ε, τη σχετική βιβλιογραφία, όπως βλέπουμε και από τον αριθμό των παραπομπών, 22.000 τέτοια πρότυπα έχουν ε, θεωρηθεί ε, prior art, όπως λέμε, το 2017 και έχει αυξηθεί η συνολική κυκλοφορία των εγγράφων αυτών κατά 2 τρίτα, κατά 60%. Και αυτό αφορά κάποιους ε, τομείς ε, κλειδιά της ε, τεχνολογίας. Επίσης χρησιμοποιούμε πληροφορίες για τα διπλώματα ευαισθητεχνίας για να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Η Κομισιόν σημειώνει στην ανακοίνωσή της για τα SCP e ότι αυτή τη στιγμή η μόνη ε, προσβάσιμη ενημέρωση για τα SCP e μπορούν, μπορεί να βρεθεί μόνο στις ε, σχετικές τράπεζες δεδομένων των SSOs. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ε, links με τις τράπεζες δεδομένων των οργανισμών αυτών για να αυξηθεί η διαφάνεια. Έχουμε ήδη αυξ... εγκαταστήσει συνέσμους με την ESPASNET όπως και τις τράπεζες ε, δεδομένων των υποβολών SCP e της ETSI για τα τηλεπικοινωνιακά πρόκυπα και της ITU. Έτσι βελτιώνουμε την διαφάνεια των SCP e μέσω μιας προσβασιμότητα που είναι φιλική προς το χρήστη, λέει ο μιλητή. και θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα στι επόμενε διαφάνειες. Πριν το κάνω αυτό όμως, θα ήθελα να σημειώσω δύο διαφορές που είναι σημαντικές στο πλαίσιο αυτό. Καταρχάς, δεν έχει κάθε οργανισμός τυποποίησης τέτοια τράπεζα δεδομένων. Η έτσι και η ITU είναι μάλλον εξαιρέσει. Δεύτερον, δεν απαιτούν από τα μέλη του την τυποποίηση να αναπτύξουν SCPs. Η έτσι έχει τέτοια υποχρέωση για τα μέλη της και διατηρεί και την ε, λεγόμενη τράπεζα δεδομένων IPR, όπου τηρούνται τα στοιχεία τα σχετικά με τα SCP. και αυτό λειτουργεί κατά αντίστοιχο παρόμοιο τρόπο για την ITU και έτσι με ένα απλό κλικ στην τράπεζα δεδομένων μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές του ESPASNET και να έχουμε σχετικές πληροφορίες για το πρότυπο. Και επομένως από εκεί και πέρα είναι ε, σχετικά εύκολο να ελέγξει κανείς το νομικό καθεστώς οποιοδήποτε ευρωπαϊκού διπλώματος και συνδεδεμένων εγγράφων. Εδώ μιλούμε για την δημοσίμηση εγγράφων ε, κατά τη ε, διάρκεια ισχύω οποιοδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ιδιοκτησίας ή χρήσης Το κοινό λοιπόν έχει πρόσβαση σε όλη αυτή την ε, πληροφορία μεταξύ των ε, τη, μέσω μάλλον της τράπεζας δεδομένων της EPO. Επίσης έχουμε το λεγόμενο ομοσπονδιακό μητρό, ομοσπονδοποιημένο είναι μητρό θα το λέγαμε, ε, όπου έχουμε πληροφορίες για την ε, ε περίοδο των 9 μηνών από τη στιγμή που έχει παραγωγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μετά από αυτό τηρούνται τα σχετικά στοιχεία στα εθνικά γραφεία, στις εθνικές υπηρεσίες ευρεσιτεχνίας. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν τα διαφερόμενη μέρη να βρουν τι έχει γίνει με ένα δίπλωμα μετά την παραχώρησή του. πολύ χρήσιμες ε, πληροφορίες μπορούν επίσης, μπορεί ε, επίσης να βρει κανείς μέσω του Global Dossier όπως το λέμε που είναι ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο ιστορικό των συνδεμένων εγγράφων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσω του Μητρώου της EPO και του ESPASNET μαζί με τα εθνικά γραφεία ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την ε, σχετική αλληλογραφία μεταξύ του υποβάλλοντα και του φορέα. Υπάρχει επίσης μηχανική ε, ε, μετάφραση για τα κινέζικα, ιαπωνικά και κορεατικά έγγραφα υποβολής. το ενιαίο μητρό Τις προστασίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία θα βοηθήσει επίσης την τραφάνεια και, για, και στην υποστήριξη και ε, προστασία των διπλωμάτων έναντι ε, νομικών προσφυγών. Στο μέλλον θα έχουμε πρόσβαση και σε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που εδώ καταλογοποιώ και προς το παρόν αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβάσιμες μέσω των ενίων σημείων. Οι πληροφορίες αυτές θα συμπεριλαμβάνονται στο μητρέο ε, της ε, Unitary Patent Protection της UPP ενώπιον του φορέα ε, επίλυσης διαφορών του ειδικού δικαστηρίου που θα επιλαμβάνεται προτού ολοκληρώσω θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε κάποιες στοιχές για τους λεγόμενους ελέγχους του ουσιώδους χαρακτήρα των SCP. Πόσο ουσιώδες, πόσο απαραίτητο δηλαδή είναι ένα SCP. E Οι οργανισμοί τυποποίησης που απαιτούν από τα μέλη τους να κοινοποιήσουν την περίπτωση ενός SCP e δεν επικυρώνουν, δεν εξακριβώνουν αν θέλετε τα συνδεδεμένα έγγραφα, απλώς αποτιμώνουν την, ε, αποτυπώνουν, διαβιβάζουν την ενημέρωση έτσι όπως την λαμβάνουν από τα μέλη τους. Το κατά πόσον είναι πραγματικά απαραίτητο ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την λειτουργία ενός προτύπου ε, εξαρτάται και από τη συζήτηση μεταξύ των μερών του υποβάλλοντα, του κατόχου του διπλώματος, του κατόχου της άδειας και δεν κρίνονται κατόπιν εξέτασης όλα τα διπλώματα SCP. E Υπάρχουν περιπτώσεις, μάλλον, οι, τα διπλώματα που ισχυρίζονται ότι είναι ουσιώδη η SCP e είναι περισσότερο από αυτό πραγματικά ε, αποφασίζεται ότι είναι κατόπιν εξέταση. Ε, σε πολλά από τα συστήματα υπάρχει μόνο η καλή πίστη του υποβάλλοντα που αποτυπώνεται στις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που θα μπορούσαν δυνητικά να είναι ουσιώδη, και τα οποία επιφέρουν και περιπλοκές στα νομικά και τεχνικά κείμενα ακόμα και για νομικούς ε, δικηγόρους που είναι γνώστες του τεχνικού αντικειμένου, λέει ο μιλητής. Όλα αυτά επίσης υπόκεινται σε τροπολογίες προκειμένου να αποφασίσει κανείς του κατά, πόσον δηλαδή ένα δίπλωμα αριστεχνίας θα κριθεί ουσιώδες SCP ή όχι και ο χαρακτήρας αυτός μπορεί και να μεταβληθεί χρονικά, συν το χρόνο. Το οποίο όμως άλλοι φορείς της αγοράς ε, το θεωρούν εμπόδιο πρόσβαση στην αγορά και ιδιαίτερα ατυχές στο πλαίσιο του διαδικτύου των ε, πραγμάτων όπου ακόμα λιγότερο πεπειραμένοι χρήστες συμμετέχουν. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τον υψηλό κίνδυνο η Κομισιόν σημειώζει ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εξακρίβωση ε, στους ελέγχους ε, του ουσιώδους χαρακτήρα των SCP και ενημέρωση των σχετικών υπηρεσιών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο περιπλοκότητας και προκλήσεων εδώ, ο αντίκτυπος επί της ανεξαρτησίας ε, των εξεταστών του ουσιώδους χαρακτήρα, του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου που θα πρέπει να διεξάγεται και εδώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι δεν έχουμε απλώς ένα είδος ελέγχου ουσιώδους χαρακτήρα. Αυτό θα μπορούσε να ε, ε, εξαρτάται από το πεδίο στο οποίο αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέχρι πολύ ενδελεχή τεχνικό, τεχνικό έλεγχο. Το, ο Ιαπωνικός φορέας ε, προσφέρει ένα είδος ελέγχου με το δικό του σύστημα hand-tie, όπως λέγεται, σχετικά με ε, προϊόντα που εξετάζεται κατά πόσον ή όχι εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αλλά από τότε που παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον Ιαπωνικό φορέα δεν έχει υψηλό δίκτυο απορρόφησης στην περσινή ετήσια συνάντηση των επικεφαλής των μεγαλύτερων οργανισμών πνευματικών δικαιωμάτων στον κόσμο, που λέγονται IP5, εξετάστηκε το θέμα αυτό και ίσως να ξαναγίνει αυτό στην φετινή ετήσια συνάντηση. Πάντως εμείς ως ΕΠΟ χαιρετίζουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην μελέτη της σκοπιμότητας που έχει ανακοινώσει η Κομισιόν θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να συνεισφέρομαι στον εντοπισμό όλων των σχετικών και απαραίτητων πτυχών και να συνεχίσουμε τη συζήτηση με το οποίο ολοκλήρωσα την ε, παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, thank you very much. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρέλιχ για την παρουσίαση. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσετε εκ μέρους μας και τον Πρόεδρο Καμπίνιος από την Επιτροπή μας. Ε, τον γνωρίζουμε εμείς και από το, το προηγούμενο πόστο του. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να θέσουμε κάποια ερωτήματα στους τρεις αυτούς πρώτους ομιλητές. Ε, ως Πρόεδρος θα καταγραφτώ τις θέσεις μου και θα θέσω ένα προφανές ερώτημα κύριοι, βλέπετε στο μέλλον να υπάρχει με, ε, ανάγκη νομοθέτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι προτεραιότητα η νομοθέτηση. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση πριν φτάσουμε στο να νομοθετήσουμε. Εάν ε, αντιμετωπίζουμε δυσκολίε σε επίπεδο διαφάνεια τα επόμενα χρόνια, ε, ενδεχομένως να χρειαστεί να υπάρξει κάποια νομική ε, απέτηση ε, για τους κατόχους των διπλωμάτων Τότε θα χρειαστούμε νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου πάντως αυτή τη στιγμή πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν όπως είπαν και οι συνάδελφοι σε επίπεδο συνεργασίας Διατάξει περί ενημέρωση. Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμε οι πληροφορίε σε ένα ίδιο τόπο. Ε, όπως είπε και η ΠΠΟ, πρέπει κανείς να ψάξει, να σκάψει για να βρει τι πληροφορίε. Και όπως είπε και ο Μάικλ, δεν δίνουν τις πληροφορίες όλες οι οργανώσεις προτύπων. Γίνονται λοιπόν πολλές προσπάθειες για να βελτιωθούν αυτά πριν φτάσουμε ε, στην νομοθεσία. Μπορεί να φτάσουμε και στην νομοθεσία κάποια στιγμή, αλλά για την ώρα υπάρχουν άλλα πράγματα να γίνουν πρώτα. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας, Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία να εξελίξει. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες η διαδικασία. Αυτά τα θέματα είχαν συζητηθεί ήδη σε επίπεδο SCP e ε, με διάφορε εμπλεκόμενε φορεί και ο Ευρωπαίο νομοθέτη έχει παίξει το ρόλο του. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει ευρεία υποστήριξη από όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Πρέπει αυτοί που εφαρμόζουν, αυτοί που είναι οι κάτοχοι των διπλωμάτων Ευρωτεχνία, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία και να τη στηρίζουν. Με την ανακοίνωση τη Κομισιόν γίνονται κάποια πρώτα βήματα, δεν είναι τα τελευταία βήματα, είναι τα πρώτα, είναι σημαντικά. Μπορεί να γίνουν και άλλα σε επίπεδο διαφάνεια, σε επίπεδο κατευθείαν γραμμή, κατευθείαν γραμμών και σαφήνεια που πρέπει να δοθεί μέσω αυτών. Νομίζω ότι πάντω πω πάμε προ σωστή κατεύθυνση. Είναι περίπλοκο. Είναι περίπλοκο διότι είναι πολλά και διάφορα τα συμφέροντα που εμπλέκονται εδώ. Ε, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί ε, τα στοιχεία τη ανακοίνωση αυτή, θα πρέπει να έχουμε περισσότερε κριτέ γραμμέ και μεγαλύτερη σαφήνεια ό,τι αφορά αυτέ τι αρχέ αξιολόγηση, το, το φραντ για το οποίο μιλάμε και για τι ε, διακρίσει βεβαίω. Ε, όχι ε, υπό τη μορφή όμως μιας νομοθεσίας, μέσω υπό μορφή μιας διαδικασίας. Επίσης ε, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος αυτών που καθορίζουν τα πρότυπα και ποιος είναι ο ρόλος των νομοθέτη, του Ευρωπαίου. Για να το πω απλά, εάν οργανώσουμε τα πράγματα στην Ευρώπη, θα έχουμε κάτι οργανωμένο για όλες τις τεχνολογίες, αλλά μόνο με στην Ευρώπη. Εάν όμως γίνει αυτό μέσω των οργανώσεων προτύπων, θα έχουμε μόνο για έναν τομέα, αλλά για όλο τον κόσμο. Σε ένα κλάδο για όλο τον κόσμο. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι η Ευρώπη εδώ δεν είναι μόνη τη, δεν είναι απομονωμένη. Και η Αμερική έχει παρεμφερή τεχνολογία και χρησιμοποιεί την, το ίντερνετ των πραγμάτων, η Κίνα, όλη η Ασία. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν στο σημείο ισορροπία. Ε, μιλάμε για εδαφικέ λύσει και μιλάμε για την Ευρώπη, ή μιλάμε για λύσει που θα αφορούν το σύνολο του κόσμου. Ε, διότι αν ο ιδιοκτήτη ενό μια. Ε, ενό διπλώματο δεν είναι ικανοποιημένο με την νομοθεσία, μπορεί να επιλέξει την Αμερική ή να επιλέξει την Κίνα. Ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να το λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ. Ε, γνωρίζετε βεβαίω το ρητό ότι ε, εφεύρει κάποιος, ε, εφευρίσκει ε, κάποιο στην Αμερική, το, το παράγει στην Κίνα και μετά το ρυθμίζουμε στην Ευρώπη νομοθετικά. Έτσι. Με καλό είναι να εφαρμοστεί και στην Ευρώπη όμως. Ε, ναι, ακούστε, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητέ μα, η ΠΠΟ θα συνεχίσει τι προσπάθειέ τη να βελτιώσει την ποιότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και να συνεισφέρει έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι να ενισχυθεί η διαφάνεια ε, για τα SCP. E θα συνεχίσουμε επίσης ε, να συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις είτε αυτές έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας με τις, ε, ε, τους οργανισμούς που παράγουν αυτά τα πρότυπα, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διαφάνεια, είτε ε, έχει να κάνει με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φώση θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορώ να συνεισφέρω και πολλά στην σημερινή αυτή συζήτηση αλλά έχω έτσι μια εντύπωση, αν κάτι κατάλαβα τέλο πάντων από όλα αυτά, διαρωτώ με αν μιλάμε σήμερα για το διαδίκτυο των πραγμάτων, για πρότυπα, για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τέλος πάντων θα πρέπει ε, να υπάρχει κάποια αξίωση ε, σε ό,τι αφορά ε, τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν σκεφτούμε σήμερα το διαδίκτυο των πραγμάτων, Πρέπει να υπάρχουν ε, πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, νομική, κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια δεδομένων και μετά πάμε στους παραγωγούς. Γιατί ε, νομίζω ότι ο πρώτος μίλησε για τη Huawei και άλλους ε, κατασκευαστές. Μπορούμε να τα δεχθούμε αυτά. Μπορούμε να κατοχυρώσουμε δίπλωμα ευρεσιτεχνία κάτι που κατά πάσα πιθανότητα είναι, προς, ε, είναι σε βάρο μα. Μπορεί να είναι καινοτομία κατοχυρώσιμη με δίπλωμα ευρεσιτεχνία, αλλά υπάρχουν παραθυράκια και πίσω πόρτες. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι υπεραπλουστευμένη ερώτησή μου, ε, η απλοϊκή, αλλά αυτό είναι το σχόλιο που μου έρχεται στο μυαλό. Ποιο θέλει να σχολιάσει, αν κάποιο θέλει να σχολιάσει. Εγώ μπορώ να κάνω ένα πρώτο σχόλιο και να συμπληρώσουν συνάδελφο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που αφορά το δίκτυο των πραγμάτων και ένα από του λόγου για του οποίου από πλευρά διπλώματων ευρεσιτεχνία ε, λέμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο. Ουσιαστικά το λέμε γιατί οι τηλεπικοινωνικέ εταιρείε είχαν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στα ε, τα πρότυπα και, τις, και τα διπλώματα. Αλλά σε λίγα χρόνια το πλυντήριο, ο καυστήρας, ε, το καλοριφέρ, όπως τρόπος που λειτουργεί το FSP, e όπως το λέμε. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι κατασκευαστές ίσως να έχουν να μιλήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα ΣΕΠ e και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συνδέονται με αυτά τα ουσιώδη πρότυπα. Είναι μεν κάτι το συναρπαστικό, αλλά γύρει και ζητήματα. Προστασία δεδομένων, για παράδειγμα, κάτι πολύ σημαντικό. Το είπατε κι εσεί. Τεχνικώ αυτό ε, μπορούμε να το διαχωρίσουμε από τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, αλλά δεν ε, υπάρχει λόγο και να μην το συμπεριλάβουμε σε μια γενική παρατήρηση και σε σχετική ε, ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένη ε, πολιτική πρόταση. Ε, δηλαδή υπάρχει ο φόβος κάποια στοιχεία να συλλέγονται, να μην έχουν έλεγχο, να πουληθούν σε τρίτους. Άρα αν θέλουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα με τα ΣΕΠ, ώστε νέες εταιρείε και ιδίω αυτές που προηγουμένως δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιούν τέτοια κατοχυρωμένη τεχνολογία, να έχουν την εμπιστοσύνη ότι μπορούν να το κάνουν και να μην φοβούνται ότι μία μέρα πριν ε, κυκλοφορεί στο προϊόν του, θα του κάνουν ασφαλιστικά μέτρα και θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε προ των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να τα δει αυτά από κοινού. Σίγουρα δεν είμαι ειδικό σε θέματα προστασία δεδομένων, αλλά δεν βλέπω και το λόγο να μην ε, τα δει υπό γενική έννοια ταυτόχρονα θα τα δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αντιδράσω στο ερώτημά σα. Είναι Πολύ θέμητο το ερώτημά σας. Είναι αλήθεια ότι η τυποποίηση είναι ένα θελοντικό σύστημα. Ε, σε ό,τι αφορά αυτούς που θέλουν να συνεισφέρουν στο πρότυπο, σε αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν και να υιοθετήσουν αυτό το πρότυπο. Από εκεί πέρα στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, όπω αυτό τη νέα προσέγγιση, δεν θα πω σε λεπτομέρειε, αλλά υπάρχει ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληρούν κάποιε ποιο, κάποια στοιχεία, κάποιε απαιτήσει. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που αναφέρει ποιε είναι οι ελάχιστε αυτές απαιτήσει. Ενσωματώνεται λοιπόν αυτό ε, στα πρότυπα που αναπτύσσουν οι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Τώρα από εκεί πέρα ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια ε, είναι επίση ε, ζητήματα τα οποία πλέον μετα... σε απαιτήσει. Υπάρχει το θέμα τη συμβατότητα ηλεκτρομαγνητική. Στο μέλλον, η κυβερνοασφάλεια, παραδείγματο χάρη, θα είναι ένα πιο σημαντικό στοιχείο. Στο τι ε, ε, θεωρούμε εμεί ω ε, βασικέ απαιτήσει. Ε, τελευταίο σχόλιο. Η διαδικασία τυποποίηση είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Όλοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει τόση ανησυχία για το hacking. Ε, το θέμα είναι ε, βέβαια άλλα πράγματα μπορεί να περάσουν από την πίσω πόρτα ό,τι φορά τις συσκευέ που θα προκύψουν. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματικού τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο τώρα, ίσως ε, για να σχολιάσει ή για να μας πει λίγο πολύ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση της ανακοίνωσης. Έχουμε 10 λεπτά. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 10 λεπτά είναι περισσότερα από όσα χρειάζομαι. Ε, δεν ήλπιζα να έχω τόσο χρόνο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που οργάνωσε αυτή την ακρόαση σήμερα, διότι πραγματικά πιστεύω ότι ε, Κάποιοι θεωρούν ότι αυτά είναι θέματα ειδικών, ε, όμως είναι πολιτικό το θέμα. Χρειάζεται στο σωστό πλαίσιο για τα πρότυπα και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γιατί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, ιδιαίτερα οι νέοι τομείς, εξαρτώνται από αυτό. Μιλάμε για IoT, αν θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές εκεί, να είμαστε στην πρώτη γραμμή, πρέπει να έχουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο στη διάθεσή μας. Και αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εκεί προσπαθούμε τουλάχιστον να συνεισφέρουμε και εμείς αυτό ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση αυτή που σας έχει απευθυνθεί ε, η προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην ανακοίνωση είναι μια προσέγγιση βήμα-βήμα σταδιακή προσέγγιση προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντές γραμμές παρουσιάζουμε την ευρωπαϊκή θέση στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και βεβαίως ε, αποφεύγουμε ευλαβικά ε, να δημιουργήσουμε στενούς κορσέδες. Θέλουμε επίσης να εφαρμόσουμε κάποιες δράσεις ε, για να εμβαθύνουμε την προσέγγιση. Είναι μια σταδιακή προσέγγιση όπως είπα. Θέλουμε μια σταδιακή δημιουργία συνένεσης γύρω από κάποιες αρχές, από κάποιες πρακτικές λύσεις που θα είναι ισορροπημένες μεταξύ τους που θα λειτουργούν για του εμπλεκόμενου φορεί, αλλά και για αυτού που εφαρμόζουν. Η ισορροπία έχει πολύ μεγάλη σημασία να λειτουργεί ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Διότι όταν μιλάμε για συνδεσιμότητα, όλε οι επιχειρήσει και οι νέε επιχειρήσει, οι startup θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποια πρότυπα. Θα πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν και στη δημιουργία των προτύπων αυτών. Όλη αυτή η κοινότητα θα πρέπει να μπορεί να έχει λύσεις που να λειτουργούν για αυτούς και να βρούμε και λύσεις οι οποίες να είναι θεκτικές στο μέλλον. Δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε τώρα ε, ε, το παρελθόν, θέλουμε το κατάλληλο πλαίσιο για το μέλλον. Διότι εκεί είναι που θα έχουμε και τα μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη ως Ευρώπη. Ε, για άλλη μια φορά τώρα, θέλω να πω ότι οι κύριοι που πήραν τον λόγο ήταν εξαιρετικοί στι παρουσιάσει του, έδωσαν κάποιε ενδείξει για το ποια είναι η προσέγγιση μα. Ε, νομίζω ότι η συνταγή τη επιτυχία ε, έχει, βασίζεται στη συνεργασία. Ε, πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων που θεσπίζουν τα πρότυπα, τα γραφεία διπλώματος ευαισθητοχνίας, στα τα εθνικά, το ευρωπαϊκό, οι πολιτικοί φορεί, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς για να βρούμε πρακτικές λύσεις Στον τομέα διαφάνειας διαφάνεια, παραδείγματο χάρη, εκεί εργαζόμαστε σκληρά και διαπιστώνουμε ότι έχει, φέρνει κάποια αποτελέσματα αυτή η προσπάθεια, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχει και ένα ζήτημα ε, ε, του να δοκιμαστούν κάποιες λύσεις ε, σε ό,τι αφορά τις άδειες. Εάν θέλουμε να βρούμε πρακτικές λύσεις ε, για, τις, για την αδειοδότηση, για την αξιολόγηση, για τους ελέγχους, κατά πόσο είναι, ένα, ε, είναι απαραίτητος, απαραίτητο δίπλωμα. Πρέπει να δοκιμαστούν πράγματα. Πολλοί συμμετέχουν στη σχετική ομάδα, πολλοί ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν επιλέξαμε 15 εμπειρογνώμονε σε πολύ ψηλό επίπεδο και ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε πολύ καλέ λύσει, ε, τι οποίε με χαρά να σα παρουσιάσω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν θα ολοκληρωθεί βέβαια η διαδικασία. Τα μελετούμε λοιπόν αυτά, τα εξετάζουμε. Γίνεται ένα brainstorming μεταξύ των διαφόρων ομάδων εμπειρογνώμονων. Ε, υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα όπω αυτό ε, για τους ελέγχους σχετικά με τον κεφαλαίωδη χαρακτήρα, τον ουσιώδη χαρακτήρα ε, ψάχνουμε λοιπόν και άλλε αυτέ γραμμέ και άλλε πρακτικέ λύσει. Τώρα σε πέδο εφαρμογή, υλοποίηση, στα πλαίσια του πακέτου μα IP, προσπαθούμε να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται και περισσότερο ε, την ε, οδηγία τη σχετική, που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία για τον κλάδο. Η αρχή τη αναλογικότητα, παραδείγματο χάρη. όταν γίνονται προσφυγέ, Εμεί συνεργαζόμαστε και με το, την δικαστική κοινότητα για να μπορούν όλα αυτά να προχωρήσουν. Βήμα-βήμα λοιπόν, σφαιρική η προσέγγιση μα. Προσπαθούμε να βρούμε πρακτικέ λύσει και ελπίζουμε ότι ω αποτέλεσμα αυτή τη εργαστηριακή δουλειά κατά κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε μέσα στο επόμενο έτος ε, ή στα δύο επόμενα έτη να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω αυτά που έχουν επιτευχθεί ω τώρα ε, πού βρίσκονται τα σημεία συμφόρηση και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και θα σκεφτούμε βεβαίω και τα επόμενα βήματα. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω και να σας πω ευχαρίστω να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους ομιλητές, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ακρόαση τη σημερινή. Προσωπικά έμαθα πολλά σήμερα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κοιμηθώ καλύτερα βέβαια μετά από αυτή την παρουσίαση, αλλά είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ακρόαση. Now the committee is going to continue in... Θα συνεχίσουμε τώρα τη συνεδρίασή μας κυκλισμένων των θυρών. Πρέπει να ζητήσω λοιπόν σε όλους όσους ε, δεν ε, έχουν θέση εδώ σε τέτοια συνεδρίαση ε, να φύγουν από την αίθουσα.